Chers collègues, Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάει η πρωινή μας συνεδρίαση. Μετά από τη συνεδρίαση θες το απόγευμα, θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας σήμερα. Σας παρακαλώ να κάνετε ησυχία. Ξεκινούμε λοιπόν σήμερα το πρωί αναφέροντας καταρχάς ότι ο κύριος Πρόεδρος, ο κύριος Κούνσταφστον, ζητά συγγνώμη, γιατί δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Θα έρθει σε μία ώρα μόλις τελειώσει η συνάντηση που έχει αυτή τη στιγμή. Και έτσι θα έρθει σε μία ώρα για το δεύτερο μέρο της πρωινής μας συνεδρίασης, δηλαδή τη συζήτηση με την Ιρλανδική Προεδρία. Θα ξεκινήσουμε με το σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης, έκθεση της κυρίας Κορνέλισεν έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας για τα δικαιώματα των γυναικών στις υποψήφιες βαλκανικές χώρες οι οποίες βρίσκονται σε φάση προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη συνεδρίαση της 3ης Οκτωβρίου του 2011 αποφασίστηκε να δοθεί αυτή η έκθεση είδης ιδίας πρωτοβουλίας στην κυρία Κορνέλισεν από την ομάδα των Πρασίνων. Είναι ένα ζήτημα εξαιρετικά σημαντικό, το ζήτημα των δικαιωμάτων των γυναικών στη Βαλκανική Χερσόνησο, στις χώρες που προσχωρούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η συζήτηση για την έκθεση αυτή σήμερα το πρωί με την κυρία Κορνέλισεν. Έχετε το λόγο, κυρία Κορνέλισεν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Το περίμενα με μεγάλη αγωνία αυτό εδώ, την ε, σημερινή μας συνεδρίαση. Πάρα πολλά χρόνια ήθελα να κάνω μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας και επιτέλους θα τη συζητήσουμε σήμερα για πρώτη φορά. Η συζήτηση θα συνεχιστεί για κάποιους μήνες από σήμερα και στο εξή θα έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε πολλές απόψεις. Ε, σας ζητώ συγγνώμη εκ μέρους των σκιωδών ε, εισηγητών που δεν μπόρεσαν να είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Το καταλαβαίνω απολύτως. Οι άλλες επιτροπές συνεδριάζουν ταυτοχρόνως σε άλλες αίθουσες και πρέπει πολλοί κόσμος να πάει αλλού για να εψηφίσει. Επισκέφθηκα τα Βαλκάνια πάρα πολλές φορές. Είμαι μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια για τις περισσότερες εκθέσεις για τις χώρες και είμαι μέλος και της Αντιπροσωπείας για την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με την πάροδο των ετών, λοιπόν, ε, νομίζω ότι μας καταθλίβει η, λίγη πρόοδος που έχει σημειωθεί. Αν όμως κανείς δει πραγματικά τα πράγματα όπως ήταν στην αρχή, πράγματι βλέπει τότε ότι η πρόοδος αυτή τελικά δεν είναι και τόσο λίγη. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις έχουν κάνει τα πάντα για να διεκδικήσουν τα δικαιώματα εθνοτικών μειονοτήτων, γυναικών, ε, λεσβιών, ομοφιλοφίλων, αμφιφιλοφίλων, φιλομεταβατικών κλπ. Νομίζω λοιπόν ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα. Οι χώρες αυτές ανήκουν στην Ευρώπη και θα πρέπει να προσχωρήσουν και η προσχώρηση αυτή θα δώσει νέα πνοή στο σεβασμό ε, των δικαιωμάτων. Εμείς ως Κοινοβούλιο καλώς ε, ε, διεκδικούμε πάντοτε το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, διότι πολύ συχνά αυτά τίθενται κατά μέρο και στρατηγούνται, Είτε μιλάμε για, την, ε, για το Κωσυφοπαίδιο, είτε μιλάμε για ε, τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Κάθε χώρα έχει άλλα προβλήματα που τελικά την κάνουν να κλείνει να θέσει τα δικαιώματα των γυναικών κατά, μέρον, κατά μέρος και γι' αυτό θέλησα να συντάξω μια τέτοια έκθεση. Αυτή τη στιγμή, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσχώρησης για τις περισσότερες χώρες, το διακύβευμα είναι η εφαρμογή. Η νομοθεσία έχει πράγματι ψηφιστεί και υιοθετηθεί. Κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των γυναικών στην νομοθεσία, αλλά οι γυναίκες δεν μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν, να τα αξιοποιήσουν τελικά στην πράξη. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις συχνά λένε ότι η χώρα μου είναι παράδεισος για τις γυναίκες επί χάρτου. Στην πράξη όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Το σχέδιο Έκθεση που παρουσιάζω βασίζεται σε μια μελέτη που θα βρείτε όλοι στο, πάνω στο θρανίο σας, στην οποία έχουν συμμετάσχει πάρα πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις, επίσημοι φορείς, μέλη των κοινοβουλίων σε αυτές τις χώρες. Εάν θέλετε ψηφιακή εκδοχή της έκθεσης αυτής, μπορεί να έρθετε σε επικοινωνία, σε επαφή με το γραφείο μου και θα σας αποστείλουμε. Στα τέλη του περασμένου Οκτωβρίου οργάνωσα ένα εργαστήριο στο Σεράγεβο με πολλούς και διαφορετικούς συνομιλητές από όλες αυτές τις χώρες ώστε να μπορέσει ο καθένας να συμβάλλει από τη μεριά του. Στο σχέδιο αυτής της έκθεσης λοιπόν προσπάθησα να επικεντρωθώ στους μηχανισμούς εφαρμογής της νομοθεσίας. Προσπάθησα να εντοπίσω κάποια γενικά ζητήματα που ισχύουν για όλες τις χώρες και προσπάθησα τέλος να αναφερθώ στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε χώρας ξεχωριστά. Με την ελπίδα ε, να ενθαρρυνθούν οι χώρες ε, ε, με αυτή την έκθεση, να νιώσουν ότι τις αφορά προσωπικά, να μην πιστέψουν οι φορείς ότι η έκθεση αφορά στις άλλες χώρες και όχι στη δική τους. Ελπίζω λοιπόν ότι με μια καλή συζήτηση θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια έκθεση χρήσιμη, αξιόλογη, που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και στη σύνταξη άλλων εκθέσεων, ώστε τελικά να μην παραμείνει νεκρό γράμμα. Ελπίζω ότι θα εγκριθεί και ότι θα εγκριθεί πριν από τον Απρίλιο, πριν τον Ιούνιο, συγγνώμη, διορθώνω. Αλλιώς αν εγκριθεί μετά την προσχώρηση της Κροατίας, η Κροατία δεν θα είναι πια υποψήφια χώρα. Άρα βλέπετε ότι έχουμε μια φυσική προθεσμία για την ε, ψήφιση της έκθεσης αυτής ε, στην Ολομέλεια. Εγώ θα κάνω το παν για να προχωρήσει το πράγμα, το πράγμα ε, και να προβληθεί η έκθεση αυτή και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων αλλά και στην αντιπροσωπεία, στον πρόεδρο της αντιπροσωπείας για την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με χαρά θα ακούσω τις παρατηρήσεις σας. Ευχαριστώ η Πρόεδρος. Ευχαριστούμε την κυρία Ισηγήτρια. Η κυρία Μποσκούγα έχει, έχει ζητήσει το λόγο και μετά η κυρία Μπάουερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλή σας μέρα. Στην ΑΦΕΤ εγώ είχα συντάξει την γνωμοδότηση για την έκθεση αυτή. Θα ήθελα καταρχήν λοιπόν να ευχαριστήσω την Μαρέια και να την συγχαρώ για την εξαιρετική έκθεσή της. Θα ε, τεθεί στην ημερήσια διάταξη και της άφετε και η ψηφοφορία θα γίνει στις 4 Μαρτίου. Συμφωνώ με την Μαρέγια Κορνέλισεν σε κάποια από τα θέματα που έχει θίξει στη δική της έκθεση. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στην εφαρμογή, διότι ωραία και καλά να έχουμε ένα κατάλογο δικαιωμάτων στο χαρτί, αλλά η πραγματική δουλειά πρέπει να γίνει από τη μεριά της εφαρμογής. Και μόνο αν μπορέσουν να ασκηθούν τα δικαιώματα αυτά στην πράξη θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο. Σημαντικό επίσης ε, είναι να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών στις χώρες αυτές και για να το πετύχουμε αυτό χρειαζόμαστε καλές στατιστικές. Αυτό είναι απαραίτητο διότι χωρίς καλές στατιστικές θα είναι πολύ πιο δύσκολο να μπορέσουμε να ελέγξουμε την κατάσταση όσον αφορά τις γυναίκες. Στην ε, γνωμοδότησή μου λοιπόν προσπάθησα να αναφέρω αυτά Επίσης, ε, τονίζω τη σημασία των μη κυβερνητικών οργανώσεων και της κοινωνία των πολιτών ε, στη διαδικασία της ε, διεύρυνσης. Σημαντικό είναι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων να παίξουν σημαντικό ρόλο τα δικαιώματα των γυναικών, εξετάζοντας την ε, έκθεση της, ε, Κομισιόν, ε, της εκθέσεις της Κομισιόν. Αυτό που βλέπει κανείς συνήθως είναι δύο παραγράφους κολλημένες στο τέλος σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών. Αλλά πρέπει να αλλάξει η κατάσταση και γι' αυτό χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα, περισσότερους πόρους για προγράμματα που στόχο έχουν τη βελτίωση της θέσης της γυναίκας. Η θυμασία της συμμετοχής ε, των γυναικών είναι σημαντική σε ε, οποιαδήποτε εγχείρημα έχει ε, να κάνει με την οικοδόμηση της δημοκρατίας. Σημαντική είναι η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, στον πολιτικό χώρο, στην οικονομία. Αυτά τονίζονται στην γνωμοδότησή μου. Τούτων λεχθέντων προσβλέπω στην συνέχεια της καλή συνεργασία με την κυρία Κορνέλησεν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μποσκιούρτη. κυρία Μπάουερ έχει το λόγο. Thank you, Elizabeth. Ευχαριστώ, Ελίζαπεθ. εκ μέρου ε, τη σκιώδου εισηγήτρια του ΕΛΚ. Ε, θα ήθελα να συγχαρώ την ε, συνάδελφό μα, την κυρία Κορνέλη, για την έκθεσή τη. Θα ήθελα δύο πράγματα να αναφέρω ε, εκ μέρους της Λίβια, της Κιόδος Συγητρίας ε, και συμφωνώ φυσικά και εγώ μαζί της. Ε, το ένα θέμα είναι η εμπορία ανθρώπων. Την προηγούμενη εβδομάδα εκδόθηκε η Παγκόσμια Έκθεση για την ε, Εμπορία Ανθρώπων που δείχνει ότι σε περιφερειακό επίπεδο ε, υπάρχει πολλή εμπορία και στην Ευρώπη συμπεριλαμβανομένης ε, και της Κεντρικής Ασίας. Η πιο σημαντική πηγή εμπορία ανθρώπων είναι τα Βαλκάνια. Πιστεύω λοιπόν ότι ε, έχει μεγάλη σημασία να τονίσουμε το θέμα της εμπορίας, διότι στην περιφέρεια αυτή γνωρίζουμε ότι εδώ και χρόνια αποτελεί πολύ σοβαρή δραστηριότητα του οργανωμένου εγκλήματος. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Συμφωνώ απόλυτα με τη Λίβια ότι πρέπει να τονίσουμε το θέμα αυτό. Το δεύτερο θέμα είναι το θέμα των Ρωμά το οποίο σε κάποιο βαθμό συνδέεται με τη, την εμπορία ανθρώπων. Γνωρίζουμε πολλές ε, υποθέσεις, πολλές περιπτώσεις ε, ε, εμπορίας ανθρώπων από το περιβάλλον των Ρωμά, αλλά το, δεν είναι η εμπορία το μόνο πρόβλημα. Έχουμε και τις πολλαπλές διακρίσεις εις βάρος των γυναικών αυτών. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω ότι παρά το γεγονός ότι είναι τόσο πλήρης η έκθεση, θα θέλαμε τουλάχιστον να τονίσουμε και αυτά τα δύο ζητήματα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Ντίτ, για αυτές τις επιπλέον πληροφορίες και για τη δική σου οπτική. Η κυρία Εύα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ως σκιώδης εισηγητή για του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτες, να ευχαριστήσω την κυρία Κορνέλισεν, που έχει αναλάβει αυτήν την σοβαρή έκθεση και του θεσμικού μηχανισμού για την αξιολόγηση των Δυτικών Βαλκανίων. Μόλι την έλαβα, δεν έχω προλάβει να τη μελετήσω, αλλά πραγματικά χαίρομαι που μα υποβάλλει μια τέτοια ποιότητα έγγραφο. Ω προ την σημερινή μα έκθεση, είναι πολύ σημαντική για να προσθεθεί στις εκθέσεις προόδου των ε, χωρών των Δυτικών Βαλκανίων που συζητούνται στην Επιτροπή ΑΦΕΤ. Για τις περισσότερες χώρες όπως αναφέρονται στην έκθεση για τα Δυτικά Βαλκάνια συμφωνώ με την εισηγήτρια για την ε, ε υλοποίηση της νομοθεσίας, την ε, ενσωμάτωση μάλλον της νομοθεσίας, η οποία δεν είναι ακόμη ολοκληρωμένη. Εξάλλου, εγώ είμαι και υπέρ του συστήματος των αποσωστώσεων που θα πρέπει μαζί με όλα τα υπόλοιπα να μεταφερθούν σωστά. Στα Δυτικά Βαλκάνια υπάρχουν ριζικέ αλλαγέ τα τελευταία χρόνια και σε αυτέ συμπεριλαμβάνονται και οι γυναίκε που είναι στην εμπροστοφυλακή τη θεσμική μεταρρύθμιση των χωρών του. Όμω, στα Δυτικά Βαλκάνια αλλάζει και η διαδικασία λήψη αποφάσεων και Αυτό βλέπουμε ότι σε καμία χώρα της Ευρώπης δεν διαφέρει γιατί καμία από τις δικές μας χώρες δεν είναι άριστη στην ε, υλοποίηση, τη σωστή υλοποίηση των αποφάσεων. Στην όλη συζήτηση θα ήθελα να επιμείνουμε λίγο περισσότερο στο θέμα της χαμηλής εκπροσώπησης των γυναικών ε, στην εργασιακή αγορά και την καταπολέμηση των ανισοτήτων των φύλων. Είναι ένα μεγάλο θέμα που συζητούμε τα τελευταία χρόνια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καλό θα ήταν λοιπόν να δοθεί έμφαση και σε αυτή την έκθεση. Τι θα μπορούσε τώρα να γίνει από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη δική μα την πλευρά. Νομίζω θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στη διαδικασία της συμπερίληψη του θέματο τη ισότητα των φύλων του mainstreaming για τις γυναίκες ε, στις περισσότερες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Νομίζω ότι θα χρειαστεί περισσότερη χρηματοδότηση για, την, για το θέμα αυτό, για το σκοπό αυτό, από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και καλό είναι να το συζητούμε στην Επιτροπή Γυναικών. Ευχαριστούμε λοιπόν την εισηγήτρια που μοιράστηκε αυτό το έγγραφο, το οποίο βρίσκω εξαιρετικό μαζί μα. Είναι πραγματικά πολύ καλή παρουσίαση τη κατάσταση των γυναικών στα Δυτικά Βαλκάνια και σχεδόν το ξέχασα. Ε, ε, διέτρεξα τα κεφάλαια αναχώρα στην έκθεση και αυτό που δεν είναι πολύ ευχάριστο είναι η κατάσταση της Κροατίας. Συζητούσα με τους παρατηρητές της ομάδας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών ε, για την Κροατία. Είδαμε μαζί την έκθεση και δεν συμφωνούν ακριβώς με όσα περιγράφει η έκθεση. Γι' αυτό ακριβώς θα φροντίσουμε να επιβάλλουμε τροπολογία σχετικά. Ακριβώς γιατί η Κροατία πρόκειται να προσχωρήσει αύριο κιόλας. Το μεγαλύτερο μέρος του κοινοτικού κεκτημένου έχει μεταφερθεί. Η Κροατία λοιπόν είναι μια χώρα στην οποία θα ήθελα να γίνουν κάποιες διορθώσεις. Ευχαριστούμε. Αλλά κυρία Κλέβα, θα μπορούσατε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένοι στις παρατηρήσεις σας για την Κροατία. Οι παρατηρητές σας δεν συμφώνησαν με τις παραγράφους όπου εκφράζονται συγχαρητήρια ή με τα εδάφια που δείχνουν ότι έχουμε υψηλότερες προσδοκίες. ακριβώς αυτό. Οι προσδοκίες μας ήταν υψηλότερες. Το μεγαλύτερο μέρος του κεκτημένου μεταφέρθηκε. Η κυβέρνηση μας της Κροατίας ήδη επεξεργάζεται την ευθυγράμμιση της νομοθεσίας της χώρας με το κοινοτικό κεκτημένο. Δεν είναι ότι δεν το λαμβάνουν υπόψη, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουν στην κατεύθυνση που έχουν ήδη, στην οποία έχουν ήδη δεσμευτεί προς την ε, προστασία της ισότητας των φύλων. Νομίζω με, τροπολογία, με σχετικές τροπολογίες θα καταστεί ακόμη σαφέστερο. Εντάξει, Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Πριν δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχω και εγώ η ίδια κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχάς, να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την κυρία Κορνέλισεν που ασχολείται με το θέμα αυτό, γιατί από τη δική μου οπτική Εάν ανοίξουν οι πόρτες της Ευρώπης για το σύνολο των χωρών των Βαλκανίων, θα πρέπει να υπάρχει παρόμοια ε, θέληση και προθυμία για την ισότητα ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς. Την ίδια προθυμία που δείχνουμε στις πολιτικές μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη δική μου αντίληψη, δεν πρέπει να έχουμε τον στόχους, αλλά να εφαρμόζουμε τις ίδιες πολιτικές και να έχουμε τις ίδιες απαιτήσει από όλους. Γι' αυτό το λόγο ακούσαμε προσοχή όσα είπατε για τη χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Νομίζω ότι πρέπει να αγωνιστούμε όχι μόνο για να φέρουμε περισσότερες γυναίκες στην αγορά εργασίας, αλλά για να υπάρχει και ισομιστία αλλά και ίση πρόσβαση σε δυνατότητε σταδιοδρομία, επαγγελματική ανέλυψη. Τρίπτυχο είναι αυτό. Ε, ισότητα γυναικο... Η εργασία των γυναικών, πρόσβαση στου μισθού και μετά στην ε, επαγγελματική ανέλυξη. Μια ολοκληρωμένη πολιτική για τους πολίτες λοιπόν σε αυτές τις χώρες που επιθυμούν να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι είναι ένα σημείο ιδιαίτερο σημαντικό και θα φροντίσω να υποβάλω σχετική τροπολογία. Δεν θα πρέπει και εμείς να υιοθετήσουμε μια εξελαχή στον αντίληψη για το τι πρέπει να περιμένουμε από τις χώρες αυτές. Όχι, θέλουμε στο επίπεδο της κοινωνίας να υπάρχει ισότητα μεταξύ των πολιτών και να βασίζεται στις δικές μας, το δικό μας επίπεδο απαιτήσεων. Σημειώνω όσα είπε και η κυρία Μπάουερ για την ανάγκη να σταθούμε ιδιαίτερως ότι γίνεται στα θέματα εμπορίας ανθρώπων, ιδίω στην εμπορία γυναικών στην γεωγραφική αυτή περιοχή. Αυτό αποτελεί ένα απόσπαστο τμήμα κατά την ε, δική μου την ε, ερμηνεία της έκθεσης αυτής. Ευχαριστώ λοιπόν την κυρία Κορνέλισεν και αν δεν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που να θέλουν το λόγο, να ακούσουμε αμέσως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρία Κάτια Ντεσάντλερ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Λέγομαι Κάτια Ντεσάντλερ. Καλύπτω την κοινωνική πολιτική και ε, θέματα απασχόλησης συμπεριλαμβανομένων θεμάτων ε, ισότητας ε, των φύλων στην Γενική Διεύθυνση για τη Διεύρυνση. Επικροτούμε την έκθεση αυτή για τα δικαιώματα των γυναικών στα Δυτικά Βαλκάνια. Επίσης, συμφωνούμε ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Είναι καλό να υιοθετούνται νόμοι αυτό το επικροτούμε, αλλά ε, βλέπουμε και εμείς από τη δική μας πλευρά ότι συχνά υστερεί η εφαρμογή. Γι' αυτό, όπως είπατε, είναι πολύ σημαντική η ευαισθητοποίηση και προσπαθήσαμε να ε, στηρίξουμε τη διαδικασία αυτή με τα δικά μας ε, προενταξιακά μέσα χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που έχουμε να ε, οργανώσουμε διάφορες εκδηλώσεις ε, και να ε, καταρτήσουμε τις αρχές των χωρών ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν σωστά την νομοθεσία που υπάρχει. Παρότι είναι σαφές ότι δεν έχουμε στις εκθέσεις πρόοδου μας πολλές παραγράφους για την ισότητα των δύο φύλων, μπορώ να πω ότι Έχουμε τακτικές επαφές με μη κυβερνητικές οργανώσεις στις χώρες αυτές, καθώς φυσικά και με τις αρχές των χωρών. Ε, και ιδιαίτερα οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις γυναικών είναι πολύ δραστήριες. Μπορώ λοιπόν να σας ενημερώσω ότι οι ομάδες που είναι αρμόδιες για τις διάφορες χώρες έχουν επαφές μαζί τους ε, για να γνωρίζουν ποια είναι η κατάσταση. Επίσης, με ικανοποίηση σημειώνω την πρόταση στο σχέδιο έκθεσης σχετικά με ε, τον διαμεσολαβητή για την ε, ισότητα των δύο φίλων στην Κροατία. Ε, καλό θα ήταν να διαδώσουμε την πρακτική αυτή. Ε, και είμαι βέβαιος ότι θα μπορεί να γίνει αυτό ε, κατά διάρκεια της βοήθειας που παρέχουμε προς άλλες χώρες ε, στη διαδικασία αυτή. Επίσης, κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με τις διάφορες χώρες όσον αφορά την Αλβανία και το, την ποσόστοση του 30%. Οι συνάδελφοί μου μου είπαν ότι αυτό μπορεί να προκαλεί κάποια σύγχυση, διότι η ποσόστοση αυτή εφαρμόζεται μόνο στα ψηφοδέλτια ε, κατά τις εκλογές. Δεν υπάρχει λοιπόν τέτοια ποσόστοση ε, όσον αφορά την αντιπροσώπευση των γυναικών ε, στην κυβέρνηση. Ίσως ε, λοιπόν ε, είναι κάπως παραπλανητική διατύπωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην έκθεση. Επίσης οι συνάδελφοί μου είπαν ότι στην Αλβανία ήδη υπάρχει επίτροπος για την ε, προστασία κατά των διακρίσεων. Η θέση δημιουργήθηκε το 2010 και ο Επίτροπος αυτός καλύπτει και θέματα ισότητας των δύο φύλων. Ίσως λοιπόν να μπορέσουμε να αναδιατυπώσουμε το σημείο 9 τονίζοντας περισσότερο ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε οι περιπτώσεις διακρίσεων λόγω ε, διακρίσεων λόγω φύλου ε, αντιμετωπίζονται επαρκώς από τον Επίτροπο. Όσον αφορά την Κροατία, μπορώ να σας ενημερώσω ότι η νομοθεσία κατά τον την αντιμετώπιση των διακρίσεων υιοθετήθηκε πέρσι το Σεπτέμβριο από την κυβέρνηση της Κροατίας. και ευθυγραμμίζεται αυτή τη στιγμή η νομοθεσία στον τομέα της ε, επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας. Ε, η Κομισιόν ε, αναλύει το, σχέδιο, το νομοσχέδιο και είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό. Περιμένουμε λοιπόν καλά νέα από την Κροατία σύντομα στο θέμα αυτό. Όσον αφορά το Μαυροβούνιο, Σημειώνω ότι γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στο κεφάλαιο 23 Δικαστικό Σώμα και Θεμελιώδη Δικαιώματα. Είναι πολύ σημαντικό το κεφάλαιο αυτό. Το σχέδιο έκθεσης ε, λοιπόν είναι ιδιαίτερα επίκαιρο, διότι όπως ίσως γνωρίζετε, οι αρχές του Μαυροβουνίου ετοιμάζουν τώρα το σχέδιο δράσης τους, ε, όπου αναφέρεται συγκεκριμένα η ισότητα των δύο φύλων. Θα πρέπει λοιπόν να υιοθετήσουν συγκεκριμένα, να αναλάβουν συγκεκριμένα βήματα για να διασφαλίσουν την ισότητα των δύο φύλων στο Μαυροβούνιο. Επίσης ε, ζητήσαμε να εφαρμόσουν μέτρα ευαισθητοποίησης και στήριξης, ιδιαίτερα όσον αφορά την απασχόληση και την ε, ε, εκπροσώπηση στην κυβέρνηση των γυναικών. Το κεφάλαιο 19, κοινωνική πολιτική και απασχόληση, μας ενδιαφέρει φυσικά επίσης όσον αφορά την ισότητα των δύο φύλων. Και μία ακόμα παρατήρηση για την Σερβία. Ήδη υπάρχουν μηχανισμοί στη Σερβία. Υπάρχει επίτροπος ε, για την ισότητα των δύο φύλων ε, και στο Υπουργείο Εργασίας υπάρχει διεύθυνση για την ισότητα των δύο φύλων. Δεν είναι λοιπόν πια απαραίτητο να δημιουργηθούν αυτοί οι μηχανισμοί, διότι ήδη υπάρχουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την Ευρωπαϊκή Επίτροπη για όλες αυτές τις διευκρινήσεις. Όπως το είπατε και εσείς, και πολύ σωστά μάλιστα, και όπως και το υπογράμμισαν πολλοί συνάδελφοι, έχουμε τις αρχές που ισχύουν, αλλά άλλη είναι η πραγματικότητα στην πράξη. Να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, διότι είδα ότι επικεντρώθηκε κυρίως ε, στο τι συμβαίνει επί τόπου. Οι αρχές που διακηρύσουμε δεν αρκούν πάντοτε. Η κυρία Κορνέλησεν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους και όλες για τις ε, πολύ λεπτομερείς και ενδελεχείς παρατηρήσεις σας. Να σχολιάσω κάποιες από αυτές, αν μου επιτρέπετε. Ορισμένοι ομιλητές μίλησαν για τη σωματεμπορία. Είναι πολύ σημαντικό να συμπεριληφθεί στην έκθεση. Να σκεφτούμε τι πρέπει να κάνει κάθε χώρα για να καταπολεμήσει αυτή τη μάστιγα. Να μην λένε μόνο οι χώρες πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι και πόσο μεγάλη ανάγκη να επιληθεί, αλλά να λένε ναι είναι μεγάλο πρόβλημα και αυτά και αυτά πρέπει να κάνουμε για να το επιλύσουμε. Ελπίζω να μου υποβληθούν τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση επικοδομητικές για να τις συμπεριλάβω κιόλα. Άλλοι μιλητέ μίλησαν για το οργανωμένο έγκλημα και χαίρομαι διότι η κυρία Χάροκα ήταν μία από τις εισηγήτριες. Νομίζω ότι θα συντάξει ένα εξαιρετικό κείμενο για την ένταξη ε, της πληθυσμιακής ομάδας των Ρωμά. Ως προς τις παρατηρήσεις της κυρίας Κλέβα ότι και χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπολείπονται ως προς την εφαρμογή ε, των κεκτημένων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πόσο δίκιο έχει. Πολύ συχνά πιστεύω ότι και για τις δικές μας χώρες μέλη θα έπρεπε να είχαμε αιτήσιες εκθέσεις προόδου. Δυστυχώς δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Βέβαια, η καθυστέρηση των υφιστάμενων χωρών μελών, ορισμένων από αυτών, δεν σημαίνει ότι πρέπει να παραγνωρίσουμε, ε, να παραγνωρίσουμε τι πρέπει να διορθωθεί και να αποκατασταθεί στις χώρες των Βαλκανίων. Τώρα, ως προς την Κροατία, προτείνω να την κρατήσουμε μέσα στην έκθεση μέχρι να ψηφιστεί, αν ψηφιστεί πριν από την προσχώρηση της Κροατίας και απλά μετά να διαγραφεί το όνομά της από την έκθεση μετά την προσχώρησή της, εάν η έκθεση τελικά ψηφιστεί αργότερα. Άλλωστε, ελπίζω ότι πολλά θα διαγραφούν από την έκθεση, γιατί πολλά ήδη θα έχουν υλοποιήσει οι χώρες αυτές τους ε, ε, αμέσως επόμενους μήνες. Μακάρι ήθε να είναι μια έκθεση όσο το δυνατόν πιο άδεια και πιο κενή. Αυτό θα σημαίνει ότι πολλά θα έχουν επιτευχθεί και δεν θα χρειάζεται να επισημανθούν στην έκθεση. Καλή πρακτική είναι ο Ombudsman στην Κροατία. Εγώ έχω δουλέψει με το γραφείο του διαμεσολαβητή αυτού τα τελευταία χρόνια, στενά. Είναι πολύ καλό. Είναι το εργαλείο που λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από όλα τα μέσα και τους μηχανισμούς. Αυτό είναι το πιο χρήσιμο. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλή, καλή πρακτική. Ως προς την Αλβανία και τις ποσοστώσεις. Σίγουρα Χρειαζόμαστε μια πιο συγκεκριμένη διατύπωση εκεί. Συμφωνώ. Να υπογραμμίσω όμως ε, το, ε, το εξής. Το κείμενο δεν λέει ότι είμαστε υπέρ των ποσοστώσεων ή απολύτως κατά αυτό, αυτών. Αυτό που λέμε στην έκθεση είναι ότι εάν μια χώρα θέλει τις αποστοστώσεις και τις έχει ενσωματώσει στην νομοθεσία της, τότε θα πρέπει να τις εφαρμόζει σωστά. Έχουμε στην Ελβανία τις ποσοστώσεις για τα ψηφοδέλτια και νομίζουν οι γυναίκες ότι τελικά 30% ε, των πολιτικών, των εκλεγμένων πολιτικών θα είναι γυναίκες. Και πόρο απέχει βέβαια η κατάσταση από το να φτάσει στο 30%. Αυτό που λέμε λοιπόν εμείς είναι ότι αν μια χώρα έχει ποσοστώσεις τότε να τις ε, εφαρμόζει και να τις ε, ε, τηρούν όλοι. Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις. Νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή έκθεση στο τέλος. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ την εισηγήτρια, κυρία Κορνέλισεν. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους σκιώδεις εισηγητές, τις σκιώδεις εισηγήτριες, τους συναδέλφους και τις συναδέλφους που πήραν το λόγο σήμερα το πρωί για ένα θέμα φλέγων για μας. Το deadline για τις για τις τροπολογίες είναι 28 Ιανουαρίου στις 5 το απόγευμα. Παρακαλώ λοιπόν να υποβάλλετε τις τροπολογίες σας μέχρι τις 28 Ιανουαρίου ε, στις 5 το απόγευμα. Στη συνέχεια, στις 18 και 19 Φεβρουαρίου του 2013 θα συζητήσουμε την έκθεση στην Επιτροπή μας. Θα την ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 20 Μαρτίου του 2013 και κατά πάσα πιθανότητα θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια του Μαΐου. Παρακαλώ λοιπόν να σημειώσετε όλοι αυτό το χρονοδιάγραμμα. Περνάμε τώρα στο δεύτερο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το σημείο 10, στρατηγική για επαρκής, ασφαλής και βιώσιμες συντάξεις. Η συντάκτρια της γνωμοδότησης στην Επιτροπή για τις Γυναίκες και την Ισότητα των Φύλων είναι η κυρία Ρεζίνα Μπάστος, την οποία ευχαριστώ για τη δουλειά της. Αρμόδια επιτροπή για την έκθεση αυτή επί της ουσίας είναι η Επιτροπή για την Απασχόληση και η κυρία Ρία Όμεν Ρούιτεν είναι η βασική εισηγήτρια. Στη συνεδρίαση της 23ης ε, Απριλίου, στη συνεδρίαση των ε, συντονιστών, αποφασίσαμε ότι θα ε, ψηφίσουμε μία γνωμοδότηση εμείς στη δική μας Επιτροπή για αυτή την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας της κυρίας Ρούιτεν. Να δώσω το λόγο στην κυρία Μπάστος. Ευχαριστώ, Ελιζαμπέτ, προεδρεύουσα της Επιτροπής μας. Στην έκθεση αυτή ε, πιστώ την προσοχή σε μια πραγματικότητα που είναι γνωστή σε όλους, την γύρανση του πληθυσμού. Η γύρανση του πληθυσμού είναι ασκεί τεράστια πίεση στα συνταξιδοτικά συστήματα και στην ε, οικονομική τους βιωσιμότητα σε όλα τα κράτη-μέλη. Για το λόγο αυτό δεν μπορούμε να αμελούμε και να παραγνωρίζουμε την κατάσταση αυτή. Θα πρέπει η προτεραιότητά μας να είναι η επαναπροσαρμογή των συνταξιδοτικών συστημάτων δεδομένων των οικονομικών και δημογραφικών εξελίξεων στην Ευρώπη. Σε αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης υπογραμμίζω τις σημαντικότερες προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες στον επαγγελματικό τους βίο και οι οποίες έχουν αρνητικές συνέπειες για την σύνταξή τους. Προτεραιότητα θα πρέπει να δώσουμε στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα απασχόλησης, σε θέματα μισθών, στην διακοπή της σταδιοδρομίας και την εργασία μερικής απασχόλησης. Επίσης, επειδή ζούμε την πρώτη δεκαετία ή τέλος πάντων μόλις τελείωσε η πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις μισθολογικές ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών. Είναι σημαντικό σε τέτοιες ε, περιπτώσεις όπως των ανισοτήτων των συντάξεων να υπογραμμιστεί προτεραιότητα, η επίγουσα ανάγκη, αυτές οι ανισότητες να εξαλειφθούν. Επιμένω λοιπόν εδώ ότι οι περίοδοι κατά τις οποίες ε, άνδρες ή γυναίκες φροντίζουν είτε τα παιδιά τους είτε άλλα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, υπόψη στον υπολογισμό των ε, συντάξεων. Να θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπέρ της δημιουργίας ενός συστήματος μονάδων για τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων, δηλαδή να συνοπολογίζονται ως ε, βαθμοί αυτά για τις συντάξεις και ανδρών και γυναικών. Ορισμένα κράτη-μέλη ήδη προβλέπουν αυτή την δυνατότητα. Επίσης, ε, τονίζω κάποια μέτρα σε σχέση με το ζήτημα αυτό των ε, συντάξεων μέτρα τα οποία πρέπει να εξασφαλίζουν μια προσέγγιση υπεύθυνη λαμβάνοντας υπόψη την πραγματικότητα των περισσότερων κρατών μελών και γι' αυτό ακριβώς ξεχωρίζουν κάποιες προτάσεις που η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συμπεριλάβει στη Λευκή Βίβλο για τις συντάξεις. Η πρώτα έχει να κάνει με την ανάγκη να συσχετιστεί η ηλικία της συνταξιδότησης με το προσδόκιμο ζωής δηλαδή να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην διαβίου μάθηση, καθώς και η συμφιλίωση του επαγγελματικού, οικογενειακού και ιδιωτικού βίου, χωρίς το οποίο ε, οι γυναίκες πάντοτε θα έχουν δυσκολίες στην συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας, ως ε, και κατά συνέπεια και στις συντάξεις τους, καθώς και στην ενεργό γύρανση. Επίσης, έμφαση δίνω στην ε, εξίσωση της ηλικίας συνταξιδότησης ανδρών και γυναικών, ώστε να βελτιωθεί και το ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας των πιο ηλικιωμένων εργαζομένων, καθώς και να διασφαλιστεί το ύψος των συντάξεών τους. Άλλη σημαντική πρόταση. Η ε, βελτίωση των συνταξιδοτικών, ε, η ανάπτυξη των συμπληρωματικών συνταξιδοτικών αποταμιεύσεων, ώστε να είναι καλύτερα τα εισοδήματα των ε, συνταξιούχων και να έχουν αξιοπρεπή ε, ζωή όταν αφήνουν τον ενεργό επαγγελματικό βίο. Τώρα, για την προθεσμία υποβολής τροπολογιών, λίγη την Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου. Αυτές είναι οι βασικές ιδέες που εκφράζονται στο σχέδιο γνωμοδότησης και ελπίζω να εγκριθεί από όλους τους ε, συναδέλφους, αφού ακούσω βέβαια τις συμβολές και τις συνεισφορές τους. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ κυρία Μπαστός. Το λόγο ζήτησε η κυρία Κλειβέτη, σχέδιση συζητήτρια για τους σοσιαλιστές και η κυρία Μπάουερ για το ΕΛΚ. Κυρία Κλειβέτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτή είναι μια από τις σημαντικότερες ε, εκθέσεις. Βέβαια, όλες οι εκθέσεις έχουν τη σημασία τους, αλλά αυτή θα έλεγα είναι από τις πλέον σημαντικές. Διότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα πρόβλημα που αφορά τους πάντες, όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Όπως βλέπουμε, από την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σαφώς υπάρχει ανησυχία για την εξέβρεση λύσης σε ένα τέτοιο πρόβλημα. Αυτό το αντιλαμβάνεται και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι φυσικά έχουμε γνώση, έχουμε εκλεγεί ως εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά ξέρουμε ότι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ετοιμαστεί και πράσινο βιβλίο και λευκή βιβλίο που εξετάζει το σχετικό ζήτημα. Επίση, ο Επίτροπο Άντορ ασχολείται επισταμένω με όλο ζήτημα. Οπότε όντω και εγώ αναγνωρίζω τη σημασία του και την ανάγκη να βρεθεί λύση. Στην έκθεση αυτή με γίνεται λόγο για επαρκή συντάξει καθώ και τη βιωσιμότητα που θα πρέπει να έχουν τα συνταξιδοτικά συστήματα. Αυτό θα πρέπει να μα απασχολεί και για το παρόν αλλά και για το μέλλον. Το πρόβλημα δεν είναι να βρεθεί η καλύτερη λύση για σήμερα, γιατί ε, όλη αυτή η διαδικασία θα βρίσκεται εν εξελίξη και για το μέλλον και είναι ένα θέμα που θα ανακύπτει διαρκώ. Δεύτερον, Λαμβάνοντας αφορμή από είπε η συγκήτρια κυρία Μπάστος, δύο παρατηρήσεις. Άλλωστε αυτός είναι και ο ρόλος της κοιόδουσης συγκήτριας. Η συνάδελφος έκανε λόγο για την πραγματικότητα της γύρανσης του πληθυσμού. Είπε ότι σήμερα αυτό αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα. Θα πρέπει να την ε, σκεφτούμε αυτή την δήλωση, διότι η σύνταξη είναι ένα δικαίωμα που κατακτά κανείς, το οποίο θεμελιώνεται στην εργασία του κατά τη διάρκεια της ζωής του. Βέβαια με τη γύρανση σημαίνει ότι οι άνθρωποι ζουν περισσότερο. Από την άλλη όμως θα πρέπει να έχουμε στο νου, κατά νου ότι η σύνταξη είναι ένα δικαίωμα. Όσοι λοιπόν καταβάλουν εισφορέ κατά τη διάρκεια του επαγγελματικού του βίου σε ένα συνταξιδοτικό σύστημα, θα πρέπει τη στιγμή που φτάνουν στην ηλικία συνταξιδότηση να έχουν μια σύνταξη, όπως λέει και ο τίτλος, επαρκή, ασφαλή και βιώσιμη. Θα συμφωνήσω λοιπόν εδώ με την εισηγήτρια. για τις ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό να το δούμε. Και ως προς τις προτάσεις μου και όλους εισηγητρίας, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και άλλα στοιχεία σε αυτόν τον κατάλογο. Βεβαίω μα απασχολούν αυτά που έθιξε και η συγγήτρια σε ό,τι αφορά τα εξαρτώμενα μέλη, αλλά θα, θα πρέπει να αναζητήσουμε λύσεις και για την ε, δουλειά στο σπίτι, το νοικοκυριό. Υπάρχει σύμβαση του Διεθνού Οργανισμού εργασία για την ε, οικιακή εργασία. Εκεί αυτού του είδους εργασία ορίζεται ως εργασία κάποιου που ε, εργάζεται εντός της οικίας του και η οποία έχει μια διάρκεια στον χρόνο, αλλά θα πρέπει να γίνεται και βάσει συγκεκριμένων προποθέσεων, ορθών προϋποθέσεων, Οι γυναίκες είναι εκείνες που καθημερινά ε, ασκούν αυτού του είδους τις δραστηριότητες, αλλά δεν αναγνωρίζεται η δουλειά τους, η συνεισφορά τους. Ο στόχος λοιπόν είναι να έχουμε υπόψη ότι οι γυναίκες κάνοντας και αυτές τις δουλειές χάνουν ένα μέρος από το δυνατό ενδυνάμει εισόδημά τους. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Είναι λοιπόν σαφές ότι θα πρέπει να αποσταλεί ένα μήνυμα προς όλες τις γυναίκες της Ευρώπης να καταλάβουν ότι ζητούμε μια λύση σε αυτό το πρόβλημα και ότι η οικιακή εργασία, το νοικοκυριό, είναι κάτι που αναγνωρίζεται, ότι είναι κάτι στο οποίο δίνουμε μια προσοχή. Ένα άλλο ζήτημα που είναι πραγματικότητα καθημερινή σε μια χώρα όπως η δική μου, η Ρουμανία, είναι ότι πολλοί πολίτε αναζητούν εργασία εκτό τη χώρα του πλέον, στο εξωτερικό. Υπάρχουν κάποια στατιστικά στοιχεία ω προ την ανεργία στην χώρα μα. Αλλά αυτό που δεν έχουμε παρακολουθήσει με τέτοια στοιχεία είναι το κατά πόσον κάποιοι που φεύγουν στο εξωτερικό μπορούν να δουλεύουν παράνομα. Τι θα γίνει με τα συνταξιδοτικά δικαιώματα των ανθρώπων αυτών. Οι γυναίκε δεν είναι προστατευμένε από τέτοιου είδου κινδύνου προφανώ, Οπότε και αυτό είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη. Θα ζητήσω από όλε τι ε, συναδέλφου να σκεφτούν τι συνταξιδοτικά συστήματα γνωρίζουν από τα διάφορα κράτη-μέλη. Να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε τα κακοσκημενά και να ανταλλάξουμε μεταξύ μας καλές πρακτικές. Θα ήταν καλό να συγκεντρώσουμε όλες τις βέλτιστες, βέλτιστες πρακτικές σε ένα κοινό σύνολο, ώστε όλοι να υποφεληθούν. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Πριν ακούσουμε την κυρία Μπάουερ, η κυρία Κονέλης αν θέλει να παρέμβει. Μήπως θα μου επιτρέψει η κυρία Μπάουερ να πάρω πρώτη το λόγο, διότι πρέπει να πάω στην ε, ΑΦΕΤ να μιλήσω για τη Μακεδονία. Θα πρέπει να είμαι πολύ, θα είμαι πολύ σύντομη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η γνωμοδότηση αυτή έχει να κάνει με κάποια πολύ σημαντικά θέματα. Οι άντρες και οι γυναίκες έχουν ε, πολύ διαφορετική ε, επαγγελματική ζωή και αυτό θα πρέπει να αντισταθμιστεί στις, ε, στα συστήματα συνταξιοδότησης προωθώντας την ισότητα. Θα ήθελα να διορθώσω το σημείο 4 ή να τροποποιήσω το σημείο 4 διότι δεν πιστεύω ότι η εξίσωση της ηλικίας συνταξιοδότησης αυτομάτως οδηγεί σε μεγαλύτερη απασχόληση των πιο ηλικιωμένων, ιδιαίτερα των γυναικών. Για να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να ε, αντιμετωπίσουμε την ε, διάκριση λόγω ηλικίας, ε, κάτι που είναι ιδιαίτερα η βάρος των πιο ηλικιωμένων γυναικών. Οι εργοδότες δεν ε, προσλαμβάνουν οι ηλικιωμένες γυναίκες και θα πρέπει να ε, ασχοληθούμε και με ε, τις δυνατότητες φύλαξης των παιδιών, διότι τώρα με την οικονομία που γίνεται λόγω των μέτρων λιτότητας οι γυναίκες ηλικίας 50-60 ετών καλούνται να φροντίσουν τα εγγόνια τους και οι άλλους συγγενείς και όσο ε, καλούνται να το κάνουν αυτό, είναι πολύ δύσκολο να παραμείνουν στην αγορά εργασία. Αυτά τα δύο ε, θέματα θα ήθελα να ε, προσθεθούν με τροπολογίε. Κατά τα άλλα, να συγχαρώ την εισηγήτρια για την γνωμοδότηση. Λυπάμαι πάρα πολύ, πρέπει να φύγω. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κυρία Κορνέλη. Κορνέλησεν, η κυρία Πάουερ, για να κλείσουμε τον κατάλογο των ομιλητών. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστώ την ε, συνάδελφο, τον κύριο Μπαστός, για την εξαιρετική της έκθεση. Πιστεύω ότι πρόκειται για ένα ζήτημα ιδιαίτερα περίπλοκο. Όλες οι προηγούμενες συνάδελφοι ουσιαστικά ενίσχυσαν την άποψή μου. Δηλαδή, οι γυναίκες θα πρέπει να μπορούν να παραμείνουν όσο το δυνατόν περισσότερο στην αγορά εργασίας και αυτό είναι αυτονόητο, διότι πέραν των γυναικών άνω των 50 ετών, μόνο το 39% βρίσκονται στην αγορά εργασίας. Πιστεύω ωστόσο ότι δεν πρέπει κανείς τη μέρα την ίδια της συνταξιοδότησης να αρχίσει να σκέφτεται πώς θα αντιμετωπίσει το θέμα των συντάξεων της συνταξιοδότησης. Όχι, πρέπει να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εκπαιδεύονται οι γυναίκες που εργάζονται, οι ηλικιωμένε γυναίκες. Θα πρέπει να επικεντρωθώ σε δύο σημεία τα οποία θα μπορούσαν να μας προβληματίσουν. Δεν θα πρέπει να καταρτήσουμε ένα κατάλογο με επιθυμίες, με, πόθ, με πόθους. Ένα μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ προέρχεται όντως από την οικιακή εργασία, από τα νοικοκυριά. Όμως Πρέπει να δούμε αν μπορούμε να διατηρήσουμε και το ισχύον συνταξιδοτικό σύστημα. Θα ήθελα τώρα να μιλήσω για την όλη προβληματική των συντάξεων σε σχέση με τα διαζύγια. και τη φροντίδα εξαρτώμενων μελών οι γυναίκες που φροντίζουν τα παιδιά τους δεν μπορούν να πάρουν ε, σύνταξη για να ασχοληθούν με αυτό το είδο τη φροντίδα. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε. Επίση, δυνατότητα μεταφορά των συνταξιδοτικών δικαιωμάτων είναι κάτι που μπορούμε να συζητήσουμε. Με αφορμή ένα συγκεκριμένο παράδειγμα στη χώρα μου, την Ουγγαρία. Το Κοινοβούλιο αποφάσισε να προβλέψει ειδικό επίδομα για τα Χριστούγεννα, ένα δώρο Χριστουγέννων. Το οποίο όμω το παίρνουν μόνο όσοι κατοικούν στην επικράτεια της χώρας. Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια διακριτική μεταχείριση. Στη Σλοβακία και όχι στην Ουγγαρία. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κινητικότητα των ε, συνταξιούχων ώστε να μην υπάρχουν μέτρα διακριτική μεταχείρισης. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Μπάουερ. Για δύο λεπτά θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε και η συγγετριά μας να κάνει την καταληκτική της παρέμβαση. Κυρία Ζαγκόρσκι, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Καταρχά να ευχαριστήσω την συγγέτρια, επειδή υποστηρίζει τα βασικά μηνύματα της Λευκής Βίβλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από τότε που δημοσιεύτηκε και νομίζω ότι έχει γίνει κάποια πρόοδο στην υλοποίηση των μέτρων έκτοτε. Τον περασμένο Μάιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με την Επιτροπή Κοινωνική Προστασία ε, υιοθέτησε έκθεση για την επάρκεια των συντάξεων, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει μια λεπτομερή ανάλυση για τι αποστάσει και τι ανισότητε των φύλων στο συνταξιδοτικό σύστημα, καθώ και την ε, ανάγκη να ληφθούν υπόψη και οι μακροχρόνιε διακοπέ στην επαγγελματική σταθερομία των ανθρώπων, λόγω τη φροντίδα των παιδιών, λόγω χάρη. Αυτό είναι ένα πρόβλημα στα συνταξιδοτικά συστήματα που υπερέχουν στα περισσότερα κράτη-μέλη. Αυτές οι διακοπές τη καριέρα μπορεί να έχουν πραγματικό αντίκτυπο στο σύνολο των συνταξιδοτικών δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζητάει αυτή τη στιγμή και με το δίκτυο των εμπειρογνωμόνων για την ισότητα των φύλων, ετοιμάζοντα μια ενδελεχή έκθεση για τι ανισότητε αυτέ λόγω του φύλου στα συνταξιδοτικά συστήματα. Αυτό συζητήθηκε στα κράτη-μέλη την περασμένη εβδομάδα. Η έκθεση αυτή ελπίζουμε να περατωθεί τους ερχόμενους μήνες. Επίσης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2012, πολλά κράτη-μέλη έλαβαν συστάσεις προκειμένου να εξισώσουν την ηλικία συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών και έκτοτε, από τότε που εγκρίθηκε η λευκη Βίπλος, δύο ακόμη κράτη-μέλη, η Πολωνία και η Σλοβενία, ενέκριναν νομοθεσία για την εξίσωση της ηλικία αυτής. Τέλος, για αυτό που είπε η κυρία Κορνέλουσεν. Ναι, να έχουμε υπόψη ότι η εξίσωση της συνταξιδοτικής ηλικία και η γενικότερη αύξησή της βεβαίως λόγω του προσδοκίμου, της επέκτασης του προσδοκίμου ζωής δεν δημιουργεί αναγκαστικά περισσότερες θέσεις εργασίας για τους ηλικιωμένους εργαζομένους, ιδίως για τις γυναίκες Γι' αυτό στη Λευκή Βίβλο ζητήσαμε μια συνολική προσέγγιση ώστε να εξισορροπηθεί ο επαγγελματικό βίωσμα και η παράτασή του με τι ε, συνταξιδοτικέ ανάγκε, ώστε να λαμβάνονται υπόψη όλα τα νέα δεδομένα. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα, Πρόεδρο. Ευχαριστώ να δώσω το λόγο στην συγκεκριά μα, την κυρία Παστό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τις συναδέλφους Κλειβέτη Κορνέλισεν, την κυρία Μπάουερ, τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όλους για τις θετικέ συνεισφορές τους για το σχέδιο γνωμοδότησης. Συμφωνούμε όλοι ότι το ζήτημα αυτό είναι άκρος επίκαιρο. Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικό από κοινωνικής και πολιτικής σκοπιάς. Έχουμε σχεδόν ε, ταυτόσιμες απόψεις Υπάρχουν αδικίε που έχουν να κάνουν με τις κοινωνικές ανισότητες, την ηλικία συνταξιδότηση, διακοπέ διακοπές της Ε, μια ποικιλία παραγόντων, οι οποίες ε, βλέπουμε να ισχύουν σε πολλά κράτη-μέλη, όπου απαιτούνται τολμηρά μέτρα, τολμηρές πολιτικές, ώστε στο μέλλον και στα συνταξιδοτικά να τηρηθεί μια στάση που να προσφέρει ασφάλεια, προβλεψιμότητα, ελπίδα για το μέλλον για τους πολίτες μας. Αυτό περιμένουν από εμά, αυτό περιμένουν από τους εκλεγμένους εκπροσώπους τους. Συμφωνούμε ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ούτε επιφύλαξη για το ότι η σύνταξη αποτελεί ένα δικαίωμα για τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες με συνεισφορές καθ' όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού του βίου. Ήδη έχουμε τη σχετική διάγνωση. Υπάρχει ανάγκη να ληφθούν μέτρα και να υιοθετηθούν προτάσεις σε επίπεδο κρατών μελών αλλά νομίζω ότι έχει φτάσει η στιγμή για να γίνουν όλα αυτά. σα ευχαριστώ όλου για την ε, συνεργασία σα και περιμένω την ε, υποβολή των τροπολογιών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Θυμίζω ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι στις 20, το μεσημέρι στις 25 Ιανουαρίου, ώστε να ψηφιστεί στην Επιτροπή Γυναικών στις 19 Φεβρουαρίου 2013 και μετά ψηφοφορία στην Επιτροπή Απασχόληση στις 21 Φεβρουαρίου. Ε, το ζήτημα αυτό θα εξεταστεί στην Ολομέλεια σε άλλη φάση. Να δώσω την Προεδρία τώρα τον πρόεδρό μας, τον κύριο Γκούσταυσον, που θα υποδεχτεί την προεδρεύουσα του Συμβουλίου της Ιρλανδίας. Να συνεχίσουμε λοιπόν τη συνεδρίασή μας. Και φτάνουμε στο σημείο 11, ανταλλαγή απόψεων με την Ιρλανδική Προεδρία. Όπως γνωρίζετε, η Ιρλανδία από το Ιανουάριο έχει αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου. Προσβλέπουμε στην ε, καλή συνεργασία με την Ιρλανδική Προεδρία. Και η ε, Επιτροπή μας επισκέφθηκε τον Νοέμβριο την ε, Ιρλανδία. Είχαμε λοιπόν τη δυνατότητα να συναντηθούμε με την Υφυπουργό κυρία Λίντς. Δύο μέρες παραμείναμε εκεί. Συζητήσαμε μια σειρά θεμάτων, μάθαμε πάρα πολλά. σχετικά με ε, την Ιρλανδική Προεδρία για το εξάμεινο αυτό. Μάθαμε όμως και για τα, την, ε, τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των δύο φύλων στην Ιρλανδία. Εκτιμήσαμε πάρα πολύ την επίσκεψή μας στην Ιρλανδία. Χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν ε, που είστε παρούσα σήμερα. Ελπίζω να έχουμε μια καλή συζήτηση. Πρώτα λοιπόν θα δώσω το λόγο στην Υφυπουργό Λίντς, Κατόπιν θα δώσω το λόγο στους ε, συντονιστές που θέλουν να πάρουν το λόγο και κατόπιν θα δώσω το λόγο σε άλλα μέλη της Επιτροπής μας. Στο τέλος θα δώσουμε τη δυνατότητα στην Υφυπουργό να απαντήσει στις ερωτήσεις. Σας καλωσορίζω λοιπόν και πάλι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε παρούσα και παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ναι, συμφωνώ ότι είχαμε πολύ επικοδομητική ε, συνάντηση το Νοέμβριο. Χάρηκα που συναντηθήκαμε σε άτυπο πλαίσιο, ώστε να μπορούμε να έχουμε ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση σχετικά με θέματα που συνδέονται με τις γυναίκες. να ομολογήσω ότι βρίσκω ότι η συνάντηση αυτή άξιζε πραγματικά τον κόπο. Η αντιπροσωπεία σας ήταν ε, αρκετά μικρή, αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ επικοδομητική η συνάντηση και νομίζω ότι δημιουργήσαμε επαφές και φιλίες ε, οι οποίες θα μας βοηθήσουν στο μέλλον, διότι νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι το θέμα των γυναικών, η θέση τους στην κοινωνία και τα θέματα ισότητας είναι πράγματα που θα ωφελήσουν όχι μόνο τα μεμονωμένα κράτη-μέλη, αλλά και το σύνολο της Ευρώπης. Κύριε Πρόεδρε, με μεγάλη ευχαρίστηση ξεκινώ την ε, σημερινή συζήτηση σχετικά με το πρόγραμμα της 7ης αυτής ε, Ιρλανδικής Προεδρίας ε, και να μιλήσω για τα δικαιώματα των γυναικών στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, κύριε Πρόεδρε, είχα μια μακρά και ευρία συζήτηση μαζί σας και με μια μικρή ομάδα των συναδέλφων σας κατά την εξερευνητική επίσκεψη στο Δουβλίνο τον Νοέμβριο. Σήμερα λοιπόν θέλουμε να διευρύνουμε τη συζήτηση αυτή ώστε να ε, συμμετάσχουν όλα τα μέλη της Επιτροπής ΦΕΜ που ε, ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των δύο φύλων. Το 2013 αποτελεί την 30η επέτειο της προσχώρησης της Ιρλανδίας στην ε, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα όταν τα έξι κράτη-μέλη γίνανε εννέα. Η τελευταία Ιρλανδική Προεδρία ε, ε είδε ε, διεύρυνση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης από 15 σε 27 κράτη-μέλη. Βλέπουμε ε, επίσης ε, την διεύρυνση, της, ε, την προσχώρηση της Κροατίας το 2013 και στο μέλλον και άλλων χωρών. Η συμμετοχή λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα είχε πολύ σημαντικό αντίκτυπο για τις γυναίκες των για τις γυναίκες της Ιρλανδίας. ενισχύθηκαν τα δικαιώματα καθώς και η οικονομική ευημερία των γυναικών. και έτσι η Ιρλανδία ε, έχει από τα καλύτερα καταρτισμένα ε, ε, σώματα εργατικού δυναμικού γυναικών και ανδρών στην Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν σημαντικούς τομείς παραγωγής τροφίμων και υπηρεσιών, κάτι που δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε πριν 30 χρόνια. Η η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσέλκυσε πολλές πολυεθνικές ε, εταιρείε ε, στη χώρα μας ε, που εξερεύνησαν διάφορες δυνατότητες. Η νομοθεσία για να αντιμετωπίσουμε την διάκριση και να προωθήσουμε την ισότητα αποτέλεσαν καλές πρακτικές. Και τώρα ενισχύεται η νομοθεσία αυτή με μια νέα δομή που θα συνδέσει τα θέματα ε, ισότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα γνωρίζετε ότι η Ιρλανδία ήταν ε, ένα από τα πρώτα θύματα της ε, οικονομικής κάμψης λόγω ιδιαίτερα της υπεθέρμανσης του τομέα οικοδομών και λόγω των, των πολλών δανείων. Ξέρουμε ότι ο αντίκτυπος ε, στα, στα δύο φύλλα διαφέρει από χώρα σε χώρα. Ε, ιδιαίτερα στην Ιρλανδία επλήγησαν οι άντρες ε, του οικοδομικού τομέα. Ε, αλλά ε, έχουν πληγεί γυναίκες και αυτό είναι κάτι που απασχολεί όλη την Ευρώπη τώρα πια η, η Ιρλανδία. Επίσης, είναι η πρώτη χώρα ε, που ανέλαβε την Προεδρία ε, υποκαθεστώς μνημονίου. Ε, Είχαμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε σημαντικές προκλήσεις τα τελευταία χρόνια, αλλά με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα αναλαμβάνουμε την Προεδρία ε, και ε, κατά την αντιμετώπιση των προκλήσεων της Ιρλανδικής Προεδρίας ε, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Ιρλανδία θα κοιτάει πέρα από τα εθνικά θέματα μας για να έχει μια ευρύτερη προοπτική όπω απαιτείται από μια επιτυχημένη Προεδρία. Κύριε Πρόεδρε, καθώ Ε, και αγαπητοί βουλευτές, θα ήθελα να πω ότι η, ε, η Ιρλανδία θα συνεργαστεί με τη Λιθουανία και την ε, Ελλάδα για να συντονίσουμε τα προγράμματα των ε, τριών προεδριών μας ε, στο θέμα της ισότητας των δύο φύλων. Ελπίζω ότι οι ε, Υπουργοί Λιθουανίας και Ελλάδα θα έρθουν στο Δουβλίνο τέλη Απριλίου για να υπογράψουν μια κοινή προκήρυξη που θέμα έχει την ανάπτυξη της θέσης απασχόλησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε τη σημασία τη ισότητας των δύο φύλων ως συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Η ισότητα δεν θα πρέπει να θεωρηθεί κόστος, θα πρέπει να αποτελεί ε, ζωτικό στοιχείο μιας ισχυρής οικονομίας ε, στην οποία συμβάλλουν όλοι οι πολίτες και από, το οποίο, από την οποία μπορούν να ωφεληθούν όλοι οι πολίτες. Ε, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Δύο Φύλων που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο το 2011 αναγνωρίζει ότι οι πολιτικέ ισότητε των δύο φύλων είναι ζωτική σημασία για την οικονομική ανάπτυξη, την ευημερία και την ανταγωνιστικότητα. Η αποτελεσματική χρήση ε, του ε, ανθρωπίνου κεφαλαίου είναι ε, σημαντικό στοιχείο για την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών. Οι αλλαγέ αυτέ έχουν επηρεάσει πολύ το πρόγραμμά μα για την ισότητα των δύο φύλων και επικεντρωνόμαστε ιδιαίτερα στην οικονομική συμμετοχή των γυναικών στην Ατζέντα 2020. Ε, χάρη στην γενναιότερη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την διοργάνωση ε, διάσκεψης στα τέλη Απριλίου. Ελπίζουμε κύριε Πρόεδρε ότι θα μπορέσετε και εσείς να συμμετάσχετε στην εκδήλωση αυτή. Θα είναι τεχνική φύση η διάσκεψη αυτή. Θέλουμε ναι, να συγκεντρώσουμε εμπειρογνώμονες σε θέματα απασχόλησης και ισότητας των δύο φύλων ε, και από τα κράτη-μέλη και από ε, χώρες υποψήφιες καθώς και από τους ε, εταίρους μας στην, στον ΕΟΧ. Θέλουμε να ανοίξουμε ένα δρόμο ώστε να βελτιστοποιήσουμε τις δυνατότητες ώστε να επιτρέψουμε στις γυναίκες της Ευρώπης να χρησιμοποιήσουν ε, το δυναμικό τους και θέλουμε να βελτιστοποιήσουμε την ε, συνεισφορά των γυναικών ε, στην οικονομική ανάπτυξη και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα, πόσο μάλλον που οι ανταγωνιστές μας στον κόσμο θεωρούνται πιο προοδευτικοί από την Ευρώπη στο θέμα αυτό. Η νέα στρατηγική απασχόληση και μια σειρά πρόσφατων δηλώσεων της Επιτροπής έχουν επικεντρωθεί στην συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία ω απαραίτητη προϋπόθεση. Εάν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να πετύχει τους στόχους της ε, για το 2020 όσον αφορά την ε, απασχόληση, πρέπει να αναλάβουμε διτή προσέγγιση. Θα πρέπει να, κοιτάξουμε, να αντιμετωπίσουμε, αλλά να κοιτάξουμε και πέρα από την παρούσα οικονομική κρίση. Για να πετύχουμε τους ε, στόχους του 2020 περί απασχόλησης, θα πρέπει να συνεργαστούμε για να βελτιώσουμε το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών επικροτούμε την ε, επικέντρωση στη συμμετοχή ε, στην αγορά εργασία των γυναικών ε, στην διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Επικροτούμε επίσης και τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης για την συμμετοχή των γυναικών στην οικονομία, ε, θέλουμε να εξετάσουμε τις περιπτώσεις γυναικών που επιλέγουν την απασχόληση, αλλά ε, να ενθαρρύνουμε και τις γυναίκες σε, σε επιχειρηματικούς ρόλους. Έχουμε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα ε, πρόθεσης της ε, γυναικείας επιχειρηματικότητας ε, στην Ιρλανδία. Θα θέλαμε να ανταλλάξουμε εμπειρίες με άλλα να ακούσουμε και να μάθουμε ένας από τον άλλον σε σε πνεύμα κοινοτικό. Αγαπητοί συνάδελφοι, παρότι δεν θα έχουμε άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ισότητας κατά τη διάρκεια Τη Ιρλανδική Προεδρίας ε, θα συναντηθούν οι Υπουργοί Απασχόλησης σε ένα άτυπο Συμβούλιο Υπουργών ΕΠΣΚΟ. Οι Υπουργοί θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ε, σε ένα εργαστήριο για την ε, ισότητα των δύο φύλων, στο οποίο θα προεδρεύσω εγώ. Όπως ανέφερα νωρίτερα, έχω ευθύνη για διάφορους τομεί στην κυβέρνηση. Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι βρίσκονται επίση εντό στι της μου και γνωρίζω ότι στην Ιρλανδία είναι έλλειπη η εκπροσώπηση των γυναικών στην αγορά εργασία. Η αποσύνδεση αυτή, ε, αυτή η μη... Ε, η έλλειψη οικονομικής ανεξαρτησίας μπορεί να οδηγήσει ε, σε προβλήματα αργότερα στη ζωή τους. Έχουμε αύξηση ε, των πιο ηλικιωμένων γυναικών στην αγορά εργασία τα τελευταία χρόνια, δηλαδή ηλικία 50 με 64 ετών. Υπάρχει ακόμα σημαντικό κενό ανάμεσα στου αριθμού ε, ανδρών και γυναικών στην ε, ηλικιακή αυτή ομάδα που είναι οικονομικά δραστήριοι. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν το σεμινάριο αυτό στο πλαίσιο τη συνάντηση των Υπουργών ΕΠΣΚΟ για να έχουμε ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και να βρούμε τρόπου να βοηθήσουμε του ηλικιωμένου ανθρώπου ε, ανθρώπους ε, να βελτιώσουν την οικονομική τους ανεξαρτησία και να αποφύγουν την φτώχεια ε, σε μεταγενέστερα στάδια τη ζωή του. Θέλουμε να υποβάλουμε σημείωμα της Προεδρίας σχετικά με το αποτέλεσμα του σεμιναρίου αυτού, καθώς και γενικά του Συμβουλίου ΕΠΣΚΟ του Ιουνίου. Και ελπίζουμε ότι συνδέοντας την ισότητα των γυναικών, την ευημερία των την ισότητα των δύο φύλων, την ευημερία των γυναικών, ε, θα μπορέσουμε να προωθήσουμε τα θέματα αυτά ε, και να τα αναλάβουν οι ε, ευρωπαϊκοί θεσμοί και στο μέλλον. Στην Ιρλανδία εκτιμούμε την δουλειά της Επιτροπής σας στο δύσκολο θέμα της βίας εις των γυναικών. Ε, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνούν όσον αφορά την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Έχουμε συνεργαστεί καλά μαζί, έχουμε ε, ε, καθιερώσει σχετικό πρόγραμμα, έχουμε το, την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας καθώς και την προστασία καθώς και την προστασία των θυμάτων εγκλημάτων. Οι έρευνες που ε, ε, έχει κάνει η ΆΙΚΑ, καθώς και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ΕΠΣΚΟ ε, του Δεκεμβρίου 2012 συμβάλλουν στην κατανόησή μας και καθοδηγούν και την πολιτική μας. Είναι επίκαιρα καθότι η βία εις των γυναικών είναι το θέμα κλειδί της 57ης συνάντησης κρατών για γυναίκες που θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο. Εγώ θα είμαι επικεφαλής της Ιρλανδικής Αντιπροσωπείας και στην Ολομέλεια θα ε, στηρίξω την ε, δουλειά του CSW ε, η 56η Σύνοδος του CSW δεν κατάφερε να υιοθετήσει συμπεράσματα. Ελπίζουμε τώρα όμως Μάλλον περιμένουμε τώρα να αντιμετωπίσουμε σημαντικές προκλήσεις, αλλά από ό,τι κατάλαβα η μόνη προηγούμενη ε, περίπτωση όπου δεν υπήρξε συμφωνία, το θέμα ήταν πάλι βία εις βάρος των γυναικών. Συμφωνούμε ότι δεν υπάρχει χώρα στην Ευρώπη, δεν υπάρχει χώρα στον κόσμο όπου ε, να μην αποτελεί σημαντικό πρόβλημα η βία εις βάρος ε, των γυναικών. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι απαραίτητο όλα τα μέλη ε, των Ηνωμένων Εθνών να συνεργαστούν στενά ώστε να έχουμε μια ε, σειρά ε, συμπερασμάτων για τη βία κατά των γυναικών. Η προετοιμασία ενός εγγράφου θέσης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησε πριν πολλούς μήνες ε, και έχουν δουλέψει πάνω σε αυτό διάφοροι εμπειρογνώμονε ε, και διπλωμάτες. Ε, πιστεύω ότι η συνεργασία αυτή θα είναι ζωτική σημασία για να έχουμε τελικά ένα οριστικό κείμενο. Και ελπίζουμε έτσι με την 57η Σύνοδο να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Ελπίζω να συμμετάσχω και σε διάφορε άλλε εκδηλώσει κατά τη διάρκεια της Προεδρία. Προεδρίας. Ε, και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ακούσουμε καλές πρακτικές. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής μου στη Νέα Υόρκη στο CSW ελπίζω να μπορέσω να μιλήσω με εκπροσώπους ε, κρατών μελών ε, και να μπορέσω να διαδώσω βέλτιστες πρακτικές. Επίσης, ελπίζω να μπορέσω να προβάλλω κάποιες από τις πρωτοβουλίες που έχουν υιοθετηθεί με ε, με την υποστήριξη της ε, Ιρλανδίας ε, στις δραστηριότητες αναπτυξιακής βοήθειάς μας που έχουν ασχοληθεί και με το θέμα της βίας εις βάρος των γυναικών. Θα μεταφέρω από όλα τα θεσμικά οργάνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Νέα Υόρκη τις ευχές για επιτυχία των διαπραγματεύσεων. Η Επιτροπή ΦΕΜ ε, νομίζω θα χαρεί που θα ακούσει ότι υπάρχει σημαντική ε, πρόοδος όσον αφορά την ε, Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας κατά τη διάρκεια των τελευταίων προεδριών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την συνάδελφό σα, ε, την κυρία Παυλόβια, για την ε, δουλειά της πάνω στο θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Εντολή ε, Προστασίας αποτελεί σημαντικό κομμάτι ενός πακέτου. Θα αναγνωρίζονται χωρίς περαιτέρω διαδικασίες οι εντολές προστασίας. Έτσι θα υπάρχει συνέχεια, κατά θα υπάρχει συνέχεια στην προστασία κατά τη μετακίνηση ανθρώπων από χώρα σε χώρα, είτε για λόγους εργασίας, είτε για λόγους σπουδών ή για άλλους λόγους. Ο ε, συνάδελφός μου ε, για τα σχετικά θέματα ε, ε, έχει δεσμευτεί να ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα αυτό και η Ιλλανδική Προεδρία σκοπεύει να οικοδομήσει πάνω στη δουλειά της Κυπριακής Προεδρίας για την υιοθέτηση θεμάτων μέτρων από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατά το πρώτο εξάμεινο του 2013. για να στηρίξουμε τα θύματα εμπορίας ε, που πολύ συχνά είναι γυναίκες. Οι Ιρλανδοί συναδελφοί μου ασχολούνται ε, με την ε, παροχή πληροφόρησης πάνω στα θέματα αυτά. Αυτό θα ε, ε, βασιστεί πάνω στην ε, τετραετή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκε πέρυσι το καλοκαίρι. Και αυτό έχει να κάνει με την οδηγία για την εμπορία ανθρώπων που πρόκειται να υιοθετηθεί στις 6 Απριλίου φέτος. Επίσης έχουμε την πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου. Ε, το θέμα αυτό είναι επίκαιρο και στις ε, πιο ανεπτυγμένε και στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Ε, ειλικρινά πιστεύω ότι απομένουν πολλά να γίνουν για να πετύχουμε ισότητα των δύο φύλων. Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω τους 12 τομείς που έχουν εντοπιστεί στην πλατφόρμα, του, πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου. Οι Προεδρίες Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναλάβει εργασίες για να ε, παρακολουθήσουν τις εργασίες στις διάφορες χώρες, στους τομείς που εντοπίστηκαν στο Πεκίνο. Ε, δείκτες για 10 από τους 12 τομείς αυτούς έχουν ήδη αναπτυχθεί και η Ιρλανδία αποφάσισε το 2011 να ετοιμάσει δείκτες ε, που έχουν να κάνουν με γυναίκες και μέσα μαζικής ενημέρωσης όσον αφορά το πρόγραμμα, στο πλαίσιο του προγράμματος για την ισότητα των δύο φύλων κατά τη διάρκεια αυτής της Προεδρίας μας. Κύριε Πρόεδρε, θα γνωρίζετε ήδη την πολύ καλή δουλειά και έρευνα που γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ισότητας των Δύο Φύλων ε, και για να υποστηρίξει την ε, πλατφόρμα του Πεκίνου, αλλά και για να προωθήσει την ισότητα των δύο φύλων. Πρέπει φυσικά να αναγνωρίσω ότι εμείς στην Ιρλανδία Ε, ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για το θέμα αυτό, καθότι η ε, απόφαση για την ε, καθιέρωση του Ινστιτούτου ήταν αποτέλεσμα της τελευταίας μας προεδρίας. Η ελευθερία λόγου, η ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία θα πρέπει να γίνονται σεβαστά συνεχώ. Ε, οι ελευθερίες αυτέ ε, αναφέρονται και γίνονται σεβαστές ε, στην πλατφόρμα του Πεκίνου. Η πλατφόρμα του Πεκίνου όμω επίση υποδεικνύει ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωση μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την ισότητα των δύο φύλων και την προώθηση του ρόλου των γυναικών όλα τα διεθνή μέσα για την ισότητα των ε, γυναικών, ε, η ΣΥΝΤΑ, ε, η πλατφόρμα του Πεκίνου, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Ισότητα των Δύο Φύλων που υπεγράφει το 2010 και η στρατηγική ισότητα των δύο φύλων της Κομισιόν τονίζουν την σημασία να πετύχουμε ισότητα των δύο φύλων κατά τη λήψη αποφάσεων. Σε σχέση με τον βασικό τομέα, ε, η πλατφόρμα του Πεκίνου ε, ε, προβλέπει ρόλο για τις γυναίκες και κατά την έλλειψη αποφάσεων, όχι μόνο στην διοίκηση επιχειρήσεων, αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης κλπ. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι πάρα πολύ ευρύ θέμα και είναι πολύ δύσκολο να το ασχοληθούμε με αυτό στο πλαίσιο μιας μόνο έρευνας. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να αναγνωρίσουμε ότι πολλά ήδη έχουν γραφεί για τα στερεότυπα των δύο φύλων και θα είναι πολύ δύσκολο ε, να έχουμε ε, ποσοτικούς δείχτες πάνω στο θέμα αυτό. Γνωρίζω την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει η ΦΕΜ πάνω σε μια σειρά θεμάτων που συνδέονται με τα στερεότυπα των δύο φύλων. Η δουλειά τη ε, Ιρλανδική Προεδρία πάνω στο θέμα αυτό θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη δικτών ε, που ε, μετρούν το ρόλο των γυναικών σε, κατά τη λήψη αποφάσεων. Έχουμε εξετάσει τουλάχιστον ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης σε κάθε χώρα και βέβαια είναι κάπως ε, περιορισμένο το εγχείρημα αυτό, ε, δεδομένου του μεγέθους ε, του δείγματος, αλλά θα έχουμε, πιστεύω, μια σαφή εικόνα σχετικά με τον ρόλο των γυναικών κατά τη λήψη αποφάσεων. Δεύτερη πτυχή της έρευνας αυτής είναι η ύπαρξη πολιτικών για την πρόθεση της ισότητας των δύο φύλων σε επιχειρήσεις μέσων μαζικής ενημέρωσης βασίζεται στον, ε, στο ρόλο των γυναικών ε, κατά τη ε, διάρκεια της λήψης αποφάσεων και πρόσφατα οι Ιδανοί συναδελφοί μας ανάπτυξαν δείκτες για το ρόλο των γυναικών στον τομέα του περιβάλλοντος στην ε, διοίκηση, διακυβέρνηση, στις πολιτικές, στην πολιτική, ε, στην ε, διπλωματία και στο δικαστικό σώμα. Εξερευνήθηκαν οι ρόλοι των γυναικών και με βάση τους τομείς αυτούς θέλουμε να παρακολουθήσουμε τις τάσεις στα κράτη-μέλη όσον αφορά τον αριθμό των γυναικών που κατέχουν θέσεις διοικητικές και ε, σκοπεύουμε να στείλουμε σχέδιο συμπερασμάτων ε, στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ. Η σχετική έκθεση θα συνοδεύει ως παράρτημα τα, συμπεράσματα του Συμβουλίου και αναμένεται να δημοσιευτεί επίσης. Μπορώ να αναφερθώ στην ε, στρατηγική επικοινωνία μας για την γνωστοποίηση πληροφοριών σε σχέση με την πλατφόρμα του Πεκίνου και να υπάρξει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για τα ζητήματα προτεραιότητα. Αυτή η α, συμπερίληψη των γυναικών στη δικασία λήψη αποφάσεων με φέρνει και σε μια άλλη προτεραιότητα τη Προεδρία. Να αρχίσουν τεχνικέ εργασίε βάσει τη ε, προσπάθεια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη στήριξή του στι αρχέ Φεβρουαρίου. Ελπίζουμε εδώ να υπάρξει σημαντική πρόοδο στο θέμα αυτό κατά τη διάρκεια τη Προεδρία μα. Αυτό το θέμα περιέχει πολλές σημαντικές προκλήσεις και έχει ήδη δημοσιοποιηθεί ιδιαίτερα πριν ε, δημοσιοποιήσει τις προτάσεις της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάποια κάτι μέλη ήδη έχουν προβλέψει ποσοστώσεις για τις γυναίκες ε, διοικητικά συμβούλια, κάποια άλλοι έχουν ε, θέσει στόχους και κάποια άλλοι κράτη, κράτη έχουν καταβάλει κάποιες προσπάθειες συμπεριλαμβανομένες της Ιρλανδίας. Βεβαίως εδώ το ποσοστό είναι ακόμη μονοψήφιο. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν ε, καταλάβει ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ισότητα των φίλων στις ε, αποφάσεις που καταρτίζουν. Εδώ θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ισότητα ανδρών και γυναικών αν θέλουμε να αντίσει οικονομία. Η διεθνή έρευνα έχει δείξει ότι οι ψυχολογικοί παράγοντες και τα επιχειρησιακά ωφέλη όπου δεν ε, υπάρχει ισότητα των φίλων βελτιστοποιεί και την δικασία λήψη αποφάσεων. Αυτό επιτρέπει στα κράτη-μέλη, αυτό ισχύει μάλλον βλέπουμε να ισχύει στα κράτη-μέλη και στην στις, ε, και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν εδώ θετικέ αποφάσεις σε σχέση με την ευαισθητοποίηση και τον καθορισμό ποσοστώσεων και στόχων. Η εκπροσώπηση των γυναικών ε, αυξάνεται λοιπόν στα συμβούλια. Όμως υπάρχουν ακόμη σημαντικές διαφορές μεταξύ του ρόλου των γυναικών στα διαφορετικά συμβούλια σε κάτι μέλη και το πώς εξελίσσονται οι όλες ε, εργασίες για την μεγαλύτερη παρουσία των γυναικών στην αλυσίδα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κάνει πιο συγκεκριμένες αποφάσεις γιατί οι ευρωπαϊκές συνθήκες είναι πολύ ε, συγκεκριμένε στους στόχους που θέτουν για την επίτευξη της ισότητας των φίλων στην απασχόληση. Στο άρθρο 157 τη συνθήκη, 157 της συνθήκη ορίζεται κάτι τέτοιο, καθώ και στο 8 τη συνθήκη για τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στοχεύει στην εξάλληψη των ανισοτήτων και την προώθηση των ισοτήτων τη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Εδώ αναγνωρίζεται η σημασία τη όλη πρωτοβουλία ε, και αυτό φάνηκε και από την ε, διοργάνωση της Κυπριακής Προεδρίας ενός γεύματος εργασίας της 6 Σεπτεμβρίου του 2012, ώστε να αρχίσει να συζητιέται το θέμα αυτό. Δεν είναι μυστικό ότι τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές απόψεις για τα θέματα αυτά. Κάποιοι θέλουν ποσοστώσεις, άλλη αυτορύθμιση. Όμως πρέπει να εργαστούμε από κοινού για να διασφαλίσουμε δίκαιη διαχείριση του θέματος αυτού και πρόοδο στον τομέα. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτείνει διαδικασία για το διορισμό ε, μελών Συμβουλίου και για σκοπούς διαφάνειας. Ωστόσο, αναζητά την ε, μη επιβολή ε, περί του άχθους σε μικρομεσές λογοχάρια επιχειρήσεις και σε κάτι μέλη που ήδη έχουν αναλάβει επιτυχημένες πρωτοβουλίες. Το Συμβούλιο πραγματικά προς το κάνει να συνεργαστεί με μεγαλύτερη επιτυχία με το Κοινοβούλιο. Ελπίζω ότι τα κράτη-μέλη θα εξεύρουν δομέ που θα επιτρέψουν την ενεργό εξέταση τη πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να καταλήξουμε σε έγκαιρη συμφωνία για ένα αμοιβαίω αποδεκτό κείμενο για την οδηγία. Κείμενο που θα ενισχύσει την ισότητα των φύλων και τι ε, αποφάσει σε επίπεδο επιχειρήσεων. Όμω, αυτό δεν πρέπει να μα οδηγεί στο να υποτιμούμε τι σοβαρέ προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ως προς την οδηγία για τις άδειες μητρότητας. Η θέση μας για το θέμα αυτό, όπως ξέρετε, η εξέταση του θέματος αυτό θα σας αδιέξατο. Εγώ ίδια ε, παρέστησα πολλές συναντήσεις όπου συζητούνταν το θέμα αυτό Ιδίω ε, μια συνάντηση στην Κρακοβία με του υπουργού ε, που ασχολούνται με θέματα ισότητα επί Πολωνική Προεδρία. Τα κάτι μέλη ε, το κατέστησαν σαφέ ότι τότε δεν μπορούσαν να δεχτούν τι βασικέ τροπολογίε του Κοινοβουλίου λόγω του κόστου και τη βιωσιμότητα στι σημερινέ οικονομικέ συνθήκε. Επίση, η προσέγγιση του Κοινοβουλίου ξεπερνούσε τις ελάχιστες προδιαγραφές και απαιτήσει για μια νέα οδηγία, αλλά και τις αρχές επικουρικότητας και αναλυκότητας. Εδώ θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ξεφύγουμε από αυτό το αδιέξοδο, διότι το αδιέξοδο αυτό έχει να κάνει με την ευελιξία που το Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να δείξει. Θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε. Όμως είναι πολύ νωρίς για να εκφράσουμε υποσχέσεις που ούτε κι εγώ ούτε κι άλλοι μπορεί να μην μπορούμε να τηρήσουμε. Ο βασικό λόγο που ήρθα σήμερα εδώ είναι για να σα παρουσιάσω το ποικίλο πρόγραμμα δραστηριοτήτων που προγραμματίζουμε κατά τη διάρκεια τη Προεδρία μα. Σε σχέση με την επίτευξη της de facto ισότητας των φύλων. Έχουμε προγραμματίσει 14 ξεχωριστέ συναντήσει και εκδηλώσει σε σχέση με θέματα ισότητας των φύλων, προκειμένου να επιτύχουμε αυτήν την φιλόδοξη δέσμευση. Ελπίζουμε να την πετύχουμε. Η Ιρλανδία είναι μια χώρα που την οδηγούν υψηλέ προσδοκίε και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα είμαστε δραστήριοι προκειμένου να καταρτήσουμε νέε πρωτοβουλίε και να προωθήσουμε την ισότητα των φύλων καθώ και τι ίσε ευκαιρίε για τι γυναίκε κατά τη διάρκεια τη Προεδρία μα. Εάν δοθούν ευκαιρίε, συνοψίζοντα, θα καλύψουμε θέματα τα οποία είναι πραγματικά ποικίλα, που έχουν να κάνουν με τι γυναίκε και τα μέσα μαζική ενημέρωση, τι γυναίκες ε, στο ρόλο τους στα διάφορα συμβούλια, τον οικονομικό τους ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οικονομική συμμετοχή των γυναικών όλων των ηλικιών. Εδώ θέλουμε να βελτιώσουμε την οικονομική τους ανεξαρτησία και να βελτιώσουμε και τη δυνατότητα της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ιλλανδική Προεδρία θα είναι φιλόδοξη στο κεντρικό ρόλο που θα δώσει στις γυναίκες, προσπαθώντας να ε, δώσουμε όθηση στην Ευρώπη και την καταπολέμηση των φαινομένων βίας κατά των γυναικών. Στην επόμενη συνάντηση του Επιτροπής για την κατάσταση των γυναικών, την 57η Σύνοδο του ΟΗΕ. Είμαι στη διάθεσή σας για να ακούσω ερωτήσεις και ελπίζω να έχουμε όχι μια, μια φιλική απλώς, αλλά επικοδομητική συνεργασία με το Κοινοβούλιο και με την τόσο ενδιαφέρουσα Επιτροπή σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Λιντ. Θα μιλήσω σου ειδικά. Eh, Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κυρία Υπουργέ, χαίρομαι διότι βρήκατε το χρόνο να έρθετε εδώ, να πάρετε το λόγο στην Επιτροπή μας η εμπειρία μου με διδάσκει ότι η Επιτροπή θα έχει πάρα πολλές ερωτήσεις να σας απευθύνει. Να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως. Να δώσω πρώτα το λόγο στους συντονιστές, μετά στα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, μετά θα δώσω το λόγο στην Υπουργό για να απαντήσει και ε, θα κινηθούμε λοιπόν ανάλογα με το μέγεθος. Η κυρία Γκαμπριέλα από το ΕΛΚ πρώτη έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα στην Επιτροπή μας. Σας ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας. Καταρχάς να σας ευχηθώ επιτυχία, κάθε επιτυχία στην υλοποίηση των στόχων σας, στόχοι που είναι μεν φιλόδοξοι αλλά όχι και ανέφικτοι. Καταρχάς λοιπόν να σας ευχηστήσω την προσοχή σε δύο λέξεις κλειδιά τις οποίες επαναλάβατε κατά κόρον στην παρέμβασή σας. Πρώτον, κοινή προσέγγιση. Δεύτερον, ανταλλαγή καλών πρακτικών. Αυτός είναι, αυτό είναι πραγματικά το ζουμί. Είναι σημαντική μεθοδολογία για να προχωρήσουμε με τους φακέλους. Χαίρομαι, διότι η Ιρλανδική Προεδρία δίνει έμφαση στη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική ανάπτυξη, το γυναικείο επιχειρήν, η γυναικεία παρουσία στην αγορά εργασίας. Είναι θέματα πολύ σημαντικά. Θα σα στηρίξουμε σε αυτά γιατί και ω Επιτροπή μα ενδιαφέρουν ιδιαιτέρω. Να σα ευχηστήσω όμω την προσοχή και σε τρία ίσονο ε, σημασία θέματα συγκριτικά με το πρώτο. Πρώτον, το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς οι διάφορες χρηματοδοτήσεις ανακλάδο και πιο συγκεκριμένα για το πρόγραμμα ισότητα των φύλων, δικαιώματα και ε, πολίτης και ηθαγένεια να μην τεθεί κατά μέρο. Θέλουμε η Ιρλανδική Προεδρία να το στηρίξει αυτό. Το επίπεδο χρηματοδότηση να παραμείνει τουλάχιστον το ίδιο για όλε αυτέ τι πρωτοβουλίε για την ισότητα των δικαιωμάτων μεταξύ ανδρών και γυναικών. Δεύτερον, Χαιρόμαστε διότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση της βίας που βιώνουν οι γυναίκες και πράγματι πρέπει να προβάλλουμε μια ισχυρή κοινή ευρωπαϊκή θέση κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το καθεστώς των γυναικών, το CSW. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να παρακολουθήσετε τα συμπεράσματα που υιοθετήθηκαν το Δεκέμβριο του 2012, ώστε να ληφθούν και μέτρα ε, για να τεθούν σε ισχύ όλες αυτές οι διατάξεις. Άλλο θέμα που μου τράβηξε την προσοχή, ως κυρίως ε, το θέμα που έχει να κάνει με την πρόταση οδηγίας της κυρίας Ρέντιν. Μιλήσατε για τεχνική δουλειά που πρέπει να γίνει. Ε, από την άλλη όμως ε, προκύπτουν διαφορετικές πρακτικές στα διάφορα κρατημέλη ως προς την οδηγία αυτή. Μπορείτε να μας ενημερώσετε περαιτέρω ποια ακριβώς τεχνική δουλειά πρέπει να γίνει για να προχωρήσει αυτή η οδηγία, ε, για να προχωρήσει αυτός ο φάκελος. Χρειαζόμαστε περισσότερη ενημέρωση νομίζω ως Επιτροπή. Και τέλος νομίζω ότι στην παρέμβασή σας ε, δεν τονίσατε αρκετά, κατά τη γνώμη μου, αυτά που συμβαίνουν εκτός Ευρώπης. Στο πλαίσιο των εξελίξεων μετά την Αραβική Άνοιξη θα πρέπει ενδεχομένω η Ιρλανδική Προεδρία να βοηθήσει, ε, να βοηθήσουμε όλοι σε αυτή την μεταβατική περίοδο, ώστε οι γυναίκες να είναι ε, παρούσες στις ομάδες διαπραγμάτευσης σε όλες αυτές τις χώρες που είναι σε μεταβατική διαδικασία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε πολλούς ομιλητές. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να ακολουθήσετε το καλό παράδειγμα της κυρίας Καπριέλ, ε, να είσαστε σύντομοι και σαφείς, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε το λόγο σας όσο γίνεται περισσότερους. Η κυρία Τόμσεν από ε, τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Εγώ μελέτησα την ιστορία των γυναικών στην Ιρλανδία και έχω δει ότι πράγματι επιτύχατε πάρα πολλά πράγματα από τότε που προσχωρήσατε μαζί με τη Δανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Πρώτου του 1973. Ίσως είναι η χώρα με τις πιο ριζικές αλλαγές στην κατάσταση των γυναικών σε όλη την Ευρώπη. Είναι, μας εμπνέει όλους το παράδειγμα των ε, Ιρλανδών γυναικών και η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στη χώρα σας. Ελπίζω λοιπόν ότι θα καταφέρουμε να οριστικοποιήσουμε όλα αυτά τα θέματα, να τα λήξουμε στο τέλος της Ιρλανδικής Προεδρίας. Εγώ θα κάνω το παν για να σας βοηθήσω προς αυτή την κατεύθυνση. Θα θέλαμε να μας στηρίξετε, όπως είπε και η προηγούμενη συνάδελφος, ε, στα τα της κατά των γυναικών. Να έχουμε δικιά μας ευρωπαϊκή οδηγία η οποία θα εκπορεύεται από ε, ψήφισμα και απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα ζητεί για κάτι τέτοιο. Τέλος, θέλω να σας ρωτήσω κάτι το οποίο δεν αναφέρατε τώρα. Στο παρελθόν όμως έχετε μιλήσει έχουν αναφερθεί κάποιες υποδείξεις για την Ιρλανδική Προεδρία και είχατε πει τότε ότι ενδεχομένως θα οργανώνεται ένα σεμινάριο για τις γυναίκες και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τα media. Είναι τεράστια πρόκληση ε, η συζήτηση για τις γυναίκες στην Ευρώπη. Όταν όμως μιλούμε για τα μέσα μαζικής επικοινωνίας τελικά και όταν υπάρχει κάλυψη, οι συμμετέχοντες είναι κατά κύριο λόγο άνδρες. Καλό θα ήταν λοιπόν να μας ε, ε, να τοποθετηθείτε για το θέμα αυτό αν έχετε την καλοσύνη. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, να δώσω το λόγο στην κυρία Παρβάνοβα, η οποία αναφέρθηκε, την οποία έφερε η κυρία Λίντς στην ομιλία σας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Υπουργό. Να σας συγχαρώ γιατί έχετε πραγματικά αναλάβει πολύ έντονη δέσμευση και έχετε προβλέψει πολύ σημαντικές ε, δράσεις ε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας. Συμφωνώ με τις συναδέλφους. Θα ήθελα και εγώ να μιλήσω για τη βία κατά των γυναικών, να ξεκινήσω από τα, από τα πιο εύκολα. Στην Επιτροπή μας ολοκληρώνουμε τον τριμηρή διάλογο για το EPO και τα θέματα αστικού δικαίου, EPO Civil, μέρος των διαπραγματεύσεων ολοκληρώθηκε κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας. Θα ολοκληρώσουμε τον τριμερή διάλογο όσο νουπο στην Επιτροπή μας και ελπίζουμε ότι η Ιρλανδική Προεδρία θα μας στηρίξει γιατί είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό για να ολοκληρωθεί η σύνταξη αυτή τη νομοθεσία και να εγκριθεί τελικά. Η κυρία Ρέντιν έχει εκφράσει ανησυχίες. Ε, πιστεύει ότι καθυστερούμε και δεν πρέπει να καθυστερούμε. Ας ε, ελπίζω ότι θα μπορέσετε να πείσετε τα κράτη-μέλη ότι πρέπει να επιταχύνουν το ρυθμό τους. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερο λόγο, ως προς το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο και τα πιο συγκεκριμένα εκάστοτε προγράμματα, το πρόγραμμα για τα δικαιώματα του πολίτη, πρόγραμμα για την ε, ενθάρρυνση και προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, πρόγραμμα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Ελπίζουμε ότι θα δεσμευθείτε ε, εντόνως και θα στηρίξετε να, το αίτημά μας να μην μειωθούν τα χρήματα που δίδονται για τέτοιου είδους δραστηριότητες και πρωτοβουλίες. Τέλος, θα έχουμε την 57η Σύνοδο της Επιτροπής για τις Γυναίκες του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, εντός ολίγου. Το Δεκέμβριο άκουσα την ομιλία του πρεσβευτή σας στα Ηνωμένα Έθνη. Άκουσα ότι η χώρα σας έχει αναλάβει ισχυρή δέσμευση και στηρίζει την επίτευξη επιτυχημένης συμφωνίας επί ενός ψηφίσματος στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Εξίσου ζωτική σημασία είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρουσιάζει συνοχή, να παρουσιάζει συνέπεια και το πιο σημαντικό είναι και το εξή άλλωστε. Αν τελικά τα Έθνη και Επιτροπή συμφωνήσουν πάνω σε ένα ψήφισμα, ότι τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα το επικυρώσει. Αυτά είπε ο πρέσβη σα και πιστεύουμε όλοι στο ηγετικό, στον ηγετικό ρόλο που θα αναλάβει η Ιρλανδική Προεδρία σε αυτούς τους κρίσιμους μήνες που βρίσκονται μπροστά μας. Ότι δηλαδή θα είστε σε θέση να δεσμευθείτε εντόνως και να εμπλέξετε με και τα άλλα κράτη-μέλη σε ακόμα πιο ισχυρή παρουσία. Ευχαριστώ κύριος Ρομέρα Ιρουέδα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τρεις είναι οι παρατηρήσεις και οι ερωτήσεις που ήθελα να κάνω. Ανισότητα, βία και απασχόληση. Πρώτον, ανισότητα και ισότητα. Το πρώτο θέμα που με ενδιαφέρει. Δεν ξέρω αν το αναφέρατε, ωστόσο είναι σημαντικό να αναφέρουμε το εξής ότι έχει μπλοκαριστεί μία από τις πιο σημαντικές οδηγίες, οι οδηγίες για την ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως θρησκευτικών ε, πιστεύω, σεξουαλικού προσανατολισμού ή αναπηριών και το καθεξής. Είναι κάτι που ε, εξετάζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γνωρίζω ότι η Ιρλανδική Προεδρία επιθυμεί να κινηθούν ταχύτερα τα πράγματα ως προς αυτό. Ε, επομένως θέτω το εξής ξεκάθαρο ερώτημα πόσες πιθανότητες έχουμε τελικά να βγει κάτι κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της Ιρλανδικής Προεδρίας. Τι πιστεύετε. Δεύτερον, ως προς το θέμα της βίας. Πρώτον, το Δάφνη. Ως Επιτροπή και γενικά το Κοινοβούλιο θέλουμε να διατηρηθεί αυτή η σήμανση Δάφνη. Να είναι ένας από τους πιο ορατούς τρόπους ε, το κοινό για τη βοήθεια που δίδουμε στα θύματα ε, της βίας. Σε ποιο σημείο βρίσκεται η κατάσταση ως προς αυτό, μπορείτε να μας πείτε. Και δεύτερον, η εξωτερική διάσταση. βιαιοπραγίες εναντίον γυναικών σε όλο τον κόσμο, θάνατοι γυναικών, ε, μέσα στη βία. Ε, μέσα σε πράξεις βίας. Οι συγκρούσεις, δηλαδή κατά τόπου σε όλο τον κόσμο, έχουν ακόμα μεγαλύτερο αντίκτυπο στις γυναίκες. Η εξωτερική διάσταση, λοιπόν, είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Όλα αυτά να μπουν εκεί. Και θα είναι ένα από τα θέματα που θα θέσουμε και στη χιλιά, άλλωστε, όταν πάμε. Και ε, αυτό είναι το δεύτερο σκέλος της δεύτερης ε, ερώτησής μου. Τρίτο τώρα, η ανισότητα η μισθολογική η οποία οφείλεται στο φύλλο. Πώς θα μειωθούν οι διαφορές στην απασχόληση μεταξύ ανδρών και γυναικών και πώς θα μειωθεί και η μισθολογική διαφορά μεταξύ των εργαζομένων ανδρών και γυναικών. Έχει αξιοποιηθεί η κρίση για να μειωθούν τελικά τα δικαιώματα των γυναικών στο να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Εγώ πιστεύω ότι πολύ συχνά χρησιμοποιείται η κρίση ως δικαιολογία για να οπισθοχωρήσουμε τελικά, να πάμε προς τα πίσω. Επομένως, ως Ιρλανδική Προεδρία, πώς θα ερμηνεύετε όλα αυτά, πώς θα αντιλαμβάνεστε όλα αυτά. Άλλωστε, έχετε και άμεσο βίωμα και άμεσες εμπειρίες με την ε, κρίση. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ξέχασα να πω στην κυρία Υπουργό ότι η κυρία Παρβάνοβα είναι από την Άλτε και ο κύριος ε, Ρωμέρα Ρουέδα είναι από τους Πρασίνους. Τέλος, η κυρία Μογάν Σαχτιέ από το ΕΛΚ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα κυρία Υπουργέ να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρέμβασή σας. Ε, θα ήθελα να σας θέσω τρεις ερωτήσεις και να σας ευχαριστήσω την προσοχή σε κάποια σημεία ε, πολύ λεπτά κατά την άποψή μας. Πρώτον, αναφέρατε ότι οι νέες γυναίκες σήμερα αποτελούν μια πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία και είναι πολύ καλά μορφωμένες και καταρτισμένες. Ωστόσο, σήμερα δυσκολεύονται ιδιαιτέρως να προσχωρήσουν, να μπουν μέσα στην αγορά εργασίας. Οι μισθοί τους είναι υπολείποτε κατά πολύ από αυτούς των ανδρών, όπως είπε ο κύριος Ρομέρα, Ρωμέβα Ιρουέδα και τελικά η σταδιοδρομία τους είναι πολύ πιο περιορισμένη και πολύ πιο επίπεδη, όχι τόσο πλούσια όσο αυτή των ανδρών πώς θα προχωρήσετε στα θέματα αυτά, πώς θα ενισχυθεί η θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας και στην οικονομία. Για να το καταφέρουμε αυτό, δεν πρέπει να το κάνουμε αποσπασματικά, θα πρέπει να ασχοληθούμε με όλα τα στοιχεία, δηλαδή και στην ένταξη στην αγορά εργασίας και στην ισότητα των μισθών και στην πρόοδο, την ανέλυξη την επαγγελματική κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας. Τι σκοπεύετε να κάνετε ως προς αυτά. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση, ο αντίκτυπος της κρίσης στις γυναίκες. Εγώ είμαι η συγγήτρια της έκθεσης ίδιας πρωτοβουλίας ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό. Δεν έχουμε και μας λείπουν απεγνωσμένα πολύ συγκεκριμένα και αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία για το θέμα αυτό. Είπε ο κύριος Ρωμέβα Ιρουέδα, έχουμε την εντύπωση ότι υποχωρούν τα κεκτημένα μας λόγω της κρίσης, τα κεκτημένα των γυναικών. Έχουμε την εντύπωση ότι οι γυναίκες ε, βρίσκονται σε ακόμα πιο ασταθή και ευπαθή θέση λόγω της κρίσης των χώρο ε, εργασίας τους, όμως δεν έχουμε συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία. Τι σκοπεύετε να κάνετε ώστε να εξαναγκαστούν τα κράτη να καταπολεμήσουν τον τον αντίκτυπο της κρίσης πιο συγκεκριμένα στις γυναίκες, ώστε να μειωθεί αυτή η διαφορά. Τρίτον, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Είναι ένας κινητήριος μοχλός αναπόδραστος, ώστε ε, να εξαλειφθούν οι διαφορές και οι ανισότητες ανδρών και γυναικών. Μας επιτρέπεται με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να εφαρμόσουμε πολιτικές για την ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας, για την επιστροφή τους στο χώρο εργασίας, για την αξιολόγηση των προσόντων και των ικανοτήτων τους. Έχουμε πάρα πολλά που μπορούμε να ε, κάνουμε χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και στη συζήτηση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο ε, τα πόδια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου τρίζουν αν θέλετε το... Είναι πάρα πολύ αποδυναμωμένα, πριονίζεται το κλαδί του. Ε, τι σκοπεύετε να κάνετε ώστε να μην υπάρξει τέτοιος κίνδυνος. Να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους που έχουν συμβάλει στη συζήτηση αυτή. Αυτά προς το παρόν ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος και εμείς σας ευχαριστούμε. Να δώσω τώρα το λόγο στην Αντιπρόεδρο κυρία Εστρέλα από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, ως εισηγήτρια για την οδηγία για την ε, γονική άδεια, καταλαβαίνω ότι είναι ένα θέμα που θα σας απασχολήσει. Μιλήσατε για ένα διέξοδο το προσπαθείτε, από το οποίο προσπαθείτε να βγείτε. Αναφερθήκατε στην δουλειά που έχει γίνει επί Πολωνικής Προεδρίας. Που ε, αποτέλεσε μια προσπάθεια να ε, ξεπλοκάρει η υπόθεση, αλλά δεν αρκούσε. Ήταν εξαιρετική η δουλειά που έγινε, αλλά δεν καταφέραμε να σημειώσουμε την επιθυμητή πρόεδρο πάνω στο θέμα αυτό. Καταλαβαίνουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάποια κράτη-μέλη. λόγω της προβληματικής οικονομικής κατάστασης. Αλλά δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να καταλάβουμε γιατί το Συμβούλιο έχει μπλοκάρει το θέμα, έχει παγώσει το θέμα. Πριν δύο χρόνια το Κοινοβούλιο υιοθέτησε την έκθεσή μου και έκτοτε, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες, το Συμβούλιο δεν έχει ακόμα φανεί πρόθυμο να ξεκινήσει έστω και άτυπο διάλογο πάνω στο θέμα αυτό. Στο Κοινοβούλιο είμαστε ευέλικτοι, ανοιχτοί απέναντι στο διάλογο και είμαστε διατεθειμένοι να συζητήσουμε το θέμα με το Συμβούλιο. Αναζητούμε λοιπόν μία διέξοδο. Το Συμβούλιο για την ώρα δεν έχει υποχωρήσει. Και εφόσον δεν υπάρξει συζήτηση στο Συμβούλιο δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τη συναπόφαση, κάθε θεσμικό όργανο, είτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε το Συμβούλιο, είτε το Ευρωκοινοβούλιο, πρέπει να, αναλάβει, να αναλαμβάνει τις ευθύνες του, να ασκεί τις αρμοδιότητές του. Έχει όμως και την υποχρέωση να σέβεται τα άλλα θεσμικά όργανα. Οπότε και να συνεργάζεται μαζί τους. Έτσι θα μπορέσουμε από κοινού να ωφελήσουμε περισσότερο τους ε, πολίτες. Κάποιες ευρωπαϊκές ενώσεις από τις πλέον αντιπροσωπευτικές, όπως το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, η Κοινωνική Πλατφόρμα, πρόσφατα ξεκίνησαν εκστρατεία ώστε να διαμηνήσουν στο Συμβούλιο ότι μία διετία είναι υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι υπερβολική περίοδος αναμονής. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι η κατάσταση θα παραμείνει σε αυτό το τέλμα. Κυρία Υπουργέ, οι προσδοκίες μας από την Ιρλανδική Προεδρία είναι υψηλές. Ελπίζουμε ότι γρήγορα θα μπορέσει να βρεθεί μία διέξοδος από αυτήν την κατάσταση. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει από το Συμβούλιο προθυμία να ξεκινήσει διάλογος. Αυτό ζητούμε μόνον από το Συμβούλιο αυτή τη στιγμή. Διάλογο για να μπορέσουμε από κοινού να εξέρουμε μια λύση ισορροπημένη η οποία να ωφελεί τις ευρωπαϊκές οικογένειες και να δίνει μια απόκριση στις ανάγκες των ευρωπαϊκών οικογενειών. Επίσης, είναι γνωστό ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει δημογραφικές προκλήσεις. Πολύ σοβαρές. Η γύρανση του πληθυσμού, τα χαμηλά ποσοστά γεννήσεων απαιτούν να ληφθούν πολιτικές αποφάσεις στήριξης της μητρότητας. Υπάρχουν πολυάριθμα επιχειρήματα, ώστε να κατανοήσει το Συμβούλιο ότι δεν πρόκειται για ένα πρόβλημα που αγγίζει απλώς τις γυναίκες. Είναι ένα πρόβλημα που αφορά τους πάντες, όλη την κοινωνία. Για το λόγο αυτό, ελπίζουμε πράγματι το Συμβούλιο να μην μας αναγκάσει το θέμα αυτό να το χρησιμοποιήσουμε ως θέμα για την προεκλογική εκστρατεία του Ευρωκοινοβουλίου το 2014. θα ήταν σαν να γνωρίζουμε ότι για μια ολόκληρη κοινοβουλευτική θητεία το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να δώσει την απαιτούμενη προσοχή σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Μας λέτε ότι υπάρχουν κάποιες προτάσεις ε, που το, το Συμβούλιο δεν μπορούσε να αποδεχτεί. Ας μας πει το Συμβούλιο ποιες είναι αυτές οι προτάσεις που δεν μπορεί να αποδεχτεί. Ας μας πει ότι είναι πρόθυμο να διαπραγματευτεί. Και από κοινού, προφανώς, θα βρούμε καλύτερες λύσεις για τους Ευρωπαίους πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι κάθε τύχη στις νέες αρμοδιότητες ε, της Προεδρίας που αναλάβατε για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ποσκούρτ από τους Σοσιαλιστές, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ για την ε, <clears throat> παρέμβασή σας. Αναφερθήκατε στην καταπολέμηση της βίας εναντίον των γυναικών. Είναι προτεραιότητα της Ιρλανδικής Προεδρίας. Το βλέπουμε άλλωστε και στο πρόγραμμα της Προεδρίας σας. Θα ήθελα όμως να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για, την, ε, για τον ακροτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Ήμασταν πολύ δραστηροί διεθνώς, εσείς ε, στην Ιρλανδία, αλλά και γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει η δέσμευση για φέτος, ώστε να υπάρξει περισσότερη δουλειά για να ε, καταπολεμηθεί αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα. Πώς ακριβώς το, έχετε περιλάβει στο πρόγραμμά σας. Θα στηρίξετε τις ευρωπαϊκές δράσεις για να δοθεί ένα τέλος στον ακροτηριασμό των γυναικείων γενετικών οργάνων. Θα τοποθετηθείτε δημοσίως ως Ιρλανδική Προεδρία καταδικάζοντας την πρακτική αυτή. Θα συμμετάσχετε στις δραστηριότητες που θα οργανωθούν ανά την Ευρώπη. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερο λόγο, οριζόντια οδηγία κατά των διακρίσεων, όπως ε, το είπε και ο κ. Ρωμέβα Ιρουέδα. Ποιες θα είναι οι συγκεκριμένες δράσεις που θα αναλάβετε ως Ιρλανδική Προεδρία για το θέμα αυτό και κυρίως ως προς το θέμα της πολλαπλής διάκρισης, των πολλαπλών διακρίσεων, όταν δηλαδή γίνονται διακρίσεις και επί τη βάση του φύλου αλλά και ε, για διάφορους άλλους λόγους. Ευχαριστώ η κυρία Κράτσα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, η υποδοχή και η ανταλλαγή απόψεων με την Υπουργό, την Αρμόδα για τα θέματα ισότητος στην αρχή της κάθε Προεδρίας είναι πολύ σημαντική για μας στιγμή και έτσι νιώθουμε και σήμερα μαζί σας. Αλλά την περίοδο αυτή αισθανόμαστε ότι έχετε μια μεγάλη πρόκληση διότι έχετε συνδέσει την ε, Προεδρία με την ε, ε, ανάγκη προώθησης της ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επιπλέον πρέπει να εξασφαλίσουμε και τους πόρους για, τα, για την υλοποίηση του, του φιλόδοξου προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Και οι γυναίκες βρίσκονται στην καρδιά αυτής της πρόκλησης και αυτού του, του σχεδίου. Αναφέρθηκαν οι συνάδελφοί μου στην ανάγκη για την επιχειρηματικότητα. Είναι κάτι που αναδεικνύεται όλο και περισσότερο έντονα σήμερα στην Ευρώπη και το, η Επιτροπή μας έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα ο ρόλος των γυναικών στην ε, δημιουργική επιχειρηματικότητα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, ε, καινοτόμες δραστηριότητες, όμως και στο ρόλο των γυναικών ως τελέχη επιχειρήσεων και αυτό είναι και σχετικό βέβαια με την πρόταση οδηγίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήθελα να σας πληροφορήσω κυρία Υπουργέ ότι το, η Επιτροπή μας έχει ασχοληθεί ήδη ένα χρόνο πριν, τον Ιούλιο του 2011, ψηφίσαμε μια έκθεση, της οποίας είχα την τιμή να είμαι που αναφέρεται ακριβώς στην προώθηση των γυναικών στο leadership των επιχειρήσεων και εκεί αναδεικνύονται και οι στόχοι που θέτουμε, τη στόχος της ποσόστοσης, της δεσμευτικής, αλλά και η πολιτική που πρέπει να έχουν οι επιχειρήσεις για να μπορούν εύκολα να αναδεικνύουν στελέχη στα ανώτατα διοικητικά όργανα και να μην χρειάζονται να γίνονται βίες παρεμβάσεις όπως από πολλούς θεωρούνται οι ποσοστώσεις. Είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε τώρα σε απάντηση με αυτή την υποδομή που ήδη έχουμε να εργαστούμε σε απάντηση της, ε, ε, της ε, πρότασης της οδηγίας που ήρθε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι πολύ σημαντικό ότι θίξατε την ανάγκη ανταλλαγής καλών πρακτικών διότι υπάρχουν καλές πρακτικές ήδη στην Ευρώπη στον τομέα της νομοθεσίας. Στόχος μας είναι η Ευρώπη να αποτελεί ένα ενιαίο χώρο και όχι να έχει δύο-τρία φωτεινά παραδείγματα, εξού και η ανάγκη της οδηγίας. Ε, και για να αντιμετωπίσουμε και όλα τα, τεχνικά θέματα, της ε, την ποικιλομορφία των δομών των επιχειρήσεων, της νομοθεσίας των επιχειρήσεων από τη μια χώρα στην άλλη. Η έκθεση που θα συντάξουμε θα είναι μαζί με την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Οπότε ήδη έχουν πάρει αυτή την πρόβλεψη ότι μια αποτελεσματική πρόταση και υλοποιήσιμη πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τα νομικά θέματα. Θέλουμε να σταθούμε ε, σε αυτό ιδιαίτερα και γι' αυτό χρειαζόμαστε και την βοήθεια της ε, Προεδρίας, ούτως ώστε να, να κατηγοροποιηθούν τα θέματα, τα τεχνικά, τα νομικά και να δούμε πώς θα ωφεληθούμε καλύτερα από την ανταλλαγή καλών πρακτικών για να προχωρήσουμε γρήγορα προς αυτή την υπόθεση. Το άλλο θέμα που θέλω να θίξω, κυρία Υπουργέ, έχει σχέση με την οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις στις γυναίκες και να τονίσω ιδιαίτερα, εκτός από την ανεργία και την ανασφάλεια στην αγορά εργασίας και την υποτίμηση και, της, ε, και του αντικρίσματος της εργασίας τους, να θέσω και το θέμα της υγείας. Η οικονομική κρίση έχει επιπτώσει στην υγεία των πολιτών, είτε αυτοί είναι άστεγοι, είτε αυτοί είναι πολίτες που δυσχεραίνονται να παρακολουθήσουν, την, να επιβλέψουν την υγεία τους, αλλά και ιδιαίτερα στις γυναίκες, διότι οι γυναίκες είναι και στον τομέα αυτά, αυτό τα πρώτα θύματα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Thank you. And now the floor Ευχαριστώ. Η κυρία Κλειβέτε από τους ε, σοσιαλιστές παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλώς ήλθατε στις Βρυξέλλες. Χαίρομαι διότι έχω την ευκαιρία να σας χαιρετήσω αλλά και να σας ξαναδώ και εσάς και τους συνεργάτες σας. Είχα την ευκαιρία να σας συνεντήσω κατά τη διάρκεια της συνάντησης της αντιπροσωπείας μας με εσάς στο Δουβλίνο. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Είμαι βέβαιη ότι θα αξιοποιήσετε στο έπακρο αυτούς τους έξι μήνες. Είστε μια γυναίκα πολύ δυνατή Άλλωστε, παρενθετικά να πω ότι ε, ήρθατε με πατερίτσε σήμερα εδώ. Ήσασταν αποφασισμένοι να έρθετε παρόλα αυτά και αυτό είναι ένα μήνυμα για την αποφασιστικότητά σας νομίζω, ένα μήνυμα στην πράξη. Και τέλος θα ήθελα να αναφέρω και το εξής. Έχουμε τρία θέματα στην ημερήσια διάταξη. Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο ή είναι σύμπτωση. Είναι όμως πολύ σημαντικά και τα τρία. Πρώτον, η ατζέντα για τις ασφαλείς, βιώσιμες και παρκείς συντάξεις. Είναι ένα θέμα που εξετάζουμε εμείς εδώ στην Επιτροπή μας και χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας πραγματικά. Γνωρίζετε την κατάσταση. Είναι φλέγον το ζήτημα αυτό. Καταρχάς αυτό. Δεύτερον, Μιλήσατε για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων που εδρεύει στο Βίλνιους της Λιθουανίας. Ελπίζω να μπορέσουμε να ψηφίσουμε την έκθεση αυτή σήμερα. Κι εγώ είμαι εισηγήτρια για το Ινστιτούτο αυτό Πολλές φωνές ακούστηκαν για να μειωθεί ο προϋπολογισμός του. Σήμερα θα ψηφίσουμε την απαλλαγή για τον προϋπολογισμό. Εγώ είμαι τελείως κατά, δεν πρέπει να υπερψηφίσουμε αυτές τις περικοπές στον προϋπολογισμό ε, του Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων. Και Τέλος, ε, έχουμε και άλλη έκθεση στην ημερήσια διάταξη, η απαλλαγή για τη διαχείριση του 2011, για το γενικό προϋπολογισμό του 2011. Ελπίζω ότι με τη βοήθειά σας ε, ως Επιτροπή δεν θα έχουμε πλέον ε, υποδείξεις και παρατηρήσεις να κάνουμε. Ελπίζω ότι δεν θα υπάρξουν δηλαδή παρατηρήσεις και υποδείξεις από το ελεγκτικό συνέδριο ως προς την προώθηση των θεμάτων και του αγώνα για την εξάλληψη των ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων. Ε, πολλοί μίλησαν για το gender budgeting και θα πρέπει να κάνουμε το πάνε έτσι ώστε και τα οικονομικά ε, να ε, κινούνται με το μέρος μας και να μας ωφελούν σε αυτόν τον αγώνα κατά πολέμους ανισοτήτων. Ευχαριστώ κυρία Μπάστος παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, να ευχηθώ κάθε τύχη για την Ιρλανδική Προεδρία. Να σας πω ότι εδώ απαριθμίσατε μια σειρά από προβλήματα που αφορούν τις γυναίκες στην Ευρώπη. Και πραγματικά δεν μπορούμε να τα αμελήσουμε. Ήθελα να επιμείνω σε τρία ζητήματα. Πρώτα απ' όλα το πελιωτές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδίως ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση του, προγράμματο του προγράμματος δικαιώματα ε, των πολιτών εδώ μας απασχολεί η καταπολέμηση της βίας που ασκείται κατά των γυναικών. Υπήρξα εισηγήτρια της έκθεσης για την αξιολόγηση του προγράμματος Δάφνη, το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 και υπήρξε συμμετοχή εξαιρετική από μη κυβερνητικέ οργανώσεις πολλών κρατομελών που γνωρίζουν ε, επισταμένως και υλοποιούν όλα αυτά τα προγράμματα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών, νεαρών γυναικών και κοριτσιών. Ε, πραγματικά έχει αποκτηθεί πολύτιμη πείρα από την ε, υλοποίηση του προγράμματος αυτού. Ήθελα λοιπόν να τονίσω ότι το Κοινοβούλιο και ιδίω η Επιτροπή μας ε, παρακολουθούν την μελλοντική χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού που πλέον καλύπτεται από το πρόγραμμα για τα δικαιώματα των πολιτών. Κυρία Υπουργέ, θα γίνει αυτή η πολιτική ε, παραχώρηση, θα φροντίσετε να υπάρξει συμβασμό ώστε να μην μειωθεί η χρηματοδότηση του προγράμματος Δάφνη και στο μέλλον. Είναι επίκαιρο το ζήτημα αυτό, διότι είναι κατεπίγουσα ανάγκη να μην μειωθεί το κονδύλι του προγράμματο αυτού. Πρέπει να έχουμε συγκεκριμένε αποδείξει ότι οι οικονομικέ και κοινωνικέ κρίσει που γνωρίζουν πολλά κράτη-μέλη δεν επιβαρύνουν ακριβώ ε, τα φαινόμενα βία. Ένα άλλο ζήτημα, κύριε Υπουργέ, έχει να κάνει με την σύνταξη και την, ε, τον συνυπολογισμό της οικιακής εργασίας. Συγκεκριμένα τις διακοπές ε, του επαγγελματικού βίου των γυναικών γιατί πρέπει να φροντίσουν τα παιδιά τους ή εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας. Εάν αυτή η οικιακή εργασία υπολογίζεται για τα δικαιώματα στη συνταξιδότηση, αυτό θα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα που περιμένουμε από την Ιρλανδική Προεδρία. Και έπειτα ένα άλλο επίκαιρο ζήτημα. Οι αρνητικές συνέπειες της οικονομικής και δημοσιονομικής και κοινωνικής κρίσης που ζουν πολλά ε, κράτη-μέλη ε, είναι κάτι που μας απασχολεί. Ε, κυρία Υπουργέ, έρχεστε από ένα κράτος μέλος που δέχεται οικονομική βοήθεια από την λεγόμενη Τρόικα το ίδιο και η δική μου χώρα, η Πορτογαλία. Οι κοινωνικές, οικονομικές και δημοσιονομικές συνέπειες της κρίσης είναι καταστρεπτικές για την κοινωνία γενικότερα, αλλά ιδιαιτέρως για τις γυναίκες, οι οποίες ουσιαστικά καταλήγουν στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό. Ήθελα λοιπόν να μου πείτε κυρία Υπουργέ, εάν η Ιρλανδική Προεδρία πρόκειται να, να, να απευθύνει συγκεκριμένες συστάσεις σε κράτη-μέλη που ε, λαμβάνουν και βρίσκονται σε καθεστώς λιτότητας. Και τώρα πραγματικά τελευταίος βουλευτής πριν μπορέσει η κυρία Υπουργός να απαντήσει στις ερωτήσεις και να κάνει τα σχολεία της, η κυρία Χάνιμπολ. Ευχαριστώ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Μία ερώτηση στην Ιρλανδία. Ξέρω ότι έχετε ένα σύνταγμα Και μεγάλο πρόβλημα με την έκδοση των, με τις εκδιδόμενες γυναίκες. Μπορείτε να μας πείτε τι κάνετε για το θέμα αυτό. Πρόεδρος, Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο για να μας πείτε τι, για να μας δώσετε τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την τελευταία ερώτηση πρώτα. Όχι, δεν έχουμε νέο νόμο για την πορνεία των γυναικών στην Ιρλανδία. Βεβαίως και έχουμε νόμο για την πορνεία, κάθε χώρα ε, έχει άλλωστε, αλλά δεν έχουμε καινούριο νόμο. Αυτό το οποίο κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Προσπαθούμε μετά από μια ευρεία διαβούλευση με όλες τις πλευρές να εξετάσουμε τον νόμο αυτό και τα ε, θέματα. Είναι πολύ δύσκολο, ε, ξέρετε, ε, να συγκεράσουμε όλες τις απόψεις. Υπάρχουν άνθρωποι που εργάζονται ε, στη βιομηχανία του σεξ και άλλοι οι οποίοι βεβαίως δεν είναι μέρος αυτού του κλάδου και δεν θέλουν καθόλου να συνομιλούν μεταξύ τους. Εμείς προσπαθούμε να ε, προσεγγίζουμε τους πάντες. Υπάρχει αυτός ο διάλογος για τα, κατά πόσο την ποινική ευθύνη θα πρέπει να την έχει ο πελάτης ή όχι. Έχουμε κάνει ευρία διαβούλευση και εξετάζουμε λοιπόν όλα αυτά τα θέματα. Αλλά δεν θα υπάρξει νέος νόμος προς το παρόν. Θα ήθελα στη συνέχεια να μιλήσω για το θέμα της κρίσης, τα οικονομικά, την οικονομία γενικότερα. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα για όλα τα κράτη-μέλη. Εμείς ως Ελλαδική Προεδρία βεβαίως εκπροσωπούμε το Συμβούλιο και όχι τόσο τη δική μας χώρα, αλλά λογικό είναι να μην μπορώ πάντοτε να διαχωρίσω αυτούς τους ρόλους. Είναι φυσικό και θεμητό άλλωστε. Οπότε ε, θα μιλήσω και για το, ε, την Ιρλανδική εμπειρία. Είμαστε δικαιούχοι λοιπόν αυτού του δανείου από την Τρόικα, το οποίο και αποπληρώνουμε. Ήμασταν η πρώτη χώρα που μπήκε σε μνημόνιο και είμαστε βεβαισμένοι ότι θα είμαστε και η πρώτη χώρα που θα βγει από το μνημόνιο. Στο βαθμό του δυνατού λοιπόν προσπαθήσαμε να προστατεύσουμε τις πιο ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες από ε, τα πιο βία χτυπήματα της κρίσης. Βεβαίως δεν μπορεί κανείς να προστατεύσει όλο το λαό από την ύφεση, αλλά προσπαθήσαμε να προστατεύσουμε τους πιο ευπαθείς και νομίζω ότι το πετύχαμε αυτό. Όλοι υποφέρουν, το γνωρίζουμε βέβαια όλοι αυτό. Ωστόσο, ε, πρέπει να εξασφαλίσουμε το εξής προς τα θέματα της απασχόλησης να μην υποφέρουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες. Αυτό θα πρέπει να είναι το κύριο μέλημά μας. Και κάθε φορά που εφαρμόζουμε διάφορα προγράμματα, τα οποία είναι και εξαιρετικά αυτά που έχουμε εμείς, όχι μόνο στην Ιρλανδία, αλλά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένας πλούτος γνώσεων και εμπειριών που πρέπει να μοιραστούμε όλοι. Και ως προς το επιχειρήν και ως προς την ενθάρρυνση των γυναικών. Πολύ συχνά τονίζω το γεγονός ότι στην Ιρλανδία εκπαιδεύουμε περισσότερο αυτούς που τελικά απασχολούμε λιγότερα. Και ε, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το επανεξετάσουμε με σοβαρότητα. Δηλαδή, όσοι επιτυγχάνουν περισσότερα στο πανεπιστημιακό κομμάτι είναι τελικά αυτοί που δεν φτάνουν στα ανώτατα κλιμάκια ε, του επαγγέλματό Επαγγελματό του. Σε ορισμένους τομεί το επιτυχάνουν ε, αυτό, σε άλλους τομεί όχι. Οι μισθολογικέ ανισότητε τώρα είναι κάτι το πολύ περίπλοκο. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται απλό. Στην ουσία όμω είναι πολύ περίπλοκο. Όταν μπαίνει κανεί σε οποιαδήποτε θέση απασχόλησης, θα πρέπει να γνωρίζει ποια είναι η μισθολογική κλίμακα την οποία θα κερδίσει. Δηλαδή κάνω αίτηση για τη χή δουλειά και η οποία αμείβεται με την χή αμοιβή πάνω κάτω. Το και η διαφορά ξεκινά μετά. Άπαξ και έχουν βρει όλη αυτή τη δουλειά στους κόλπους του, του ίδιου χώρου εργασίας. Εκεί υπάρχουν οι μισθολογικές ανισότητες. Πώς θα καλύψουμε λοιπόν αυτό το κενό οι εργοδότες να είναι ενημερωμένοι και να ε, είναι πεπισμένοι να πούν ότι και να πιστούν στο ότι δεν πρόκειται να εφαρμόσουν μισθολογικές ανισότητες ακριβώς για να πάρουν τα καλύτερα από τους εργαζόμενούς τους, τους απασχολούμενούς τους. Πιστεύω ακραδάντως ότι αν κάτι καλά η Ευρώπη είναι ότι είναι το εξής. Όταν και αν αποφασίζουμε ως Ευρώπη κάτι να το προωθήσουμε, τότε πράγματι το προωθούμε και το κάνουμε καλά. Και πρέπει να δούμε πού είναι εφικτό να προχωρήσουμε. Κάθε Προεδρία έχει στη διάθεσή της μόνο έξι μήνες. Έξι μήνες και προχωρεί το φάκελο όσο μπορεί, λίγο-λίγο κάθε φορά. Ε, βασικό μας μέλημα είναι να κινείται ο φάκελος προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό θα πρέπει να μας ενδιαφέρει. Και γι' αυτό το ανέφερα και σήμερα το πρωί πολύ και διαφορετικοί, με συμβούλευσαν πολλά και διαφορετικά πράγματα για το κατά πόσο θα έπρεπε να αναφερθώ στην οδηγία για την άδεια μητρότητα. Οι μισοί μου έλεγαν μην το αναφέρεις. Άλλοι μου έλεγαν να το αναφέρεις γιατί αν δεν το αναφέρεις κάποιο βουλευτής θα το αναφέρει. Τα γνωρίζετε αυτά στην πολιτική συμβαίνουν. Αποφασίσαμε λοιπόν το εξή. Η Ευρώπη προχωράει προς τα εμπρό και θα πρέπει να μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο και στο θέμα αυτό. Αλλά θα το προσογγίσουμε, θα το αναλάβουμε μόνο εάν πιστούμε ότι πράγματι υπάρχει βούληση. Βούληση συνεργασίας. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το προχωρήσουμε. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε. Και υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο. Νομίζω ότι θα έπρεπε Νομίζω ότι αν υπάρχει βούληση πραγματική συνεργασίας, τότε θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε. Και με τις συνομιλίες, με την επικοινωνία, κατά πάσα πιθανότητα θα βρεθεί λύση. Ε, υπάρχει επικουρικότητα, υπάρχουν οι ευθύνες των κρατών μελών. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά. Και είναι και εξαιρετικά σημαντικά για εμάς στην Ιρλανδία, δεδομένου του μικρού μεγέθους της χώρας μας και σε μεγάλο βαθμό λόγω και της απόστασης της γεωγραφικής που μας χωρίζει από την ε, Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Επομένως, ε, ε, έχουμε πλήρη συνείδηση ότι οι χώρες μπορεί να έχουν ανάγκη να καθορίζουν τη μοίρα τους σε μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, αν υπάρχει βούληση συνεργασίας θα πρέπει να προχωρήσουμε αυτό το φάκελο και δεν θα ασχοληθούμε με αυτό το φάκελο αν δεν πιστούμε ότι υπάρχει πραγματική βούληση συνεργασίας. Άλλες χώρες θα πάνε εξαιρετικά καλά ως προς το ζήτημα αυτό, άλλες χώρες δεν είναι τόσο ανεπτυγμένες. Θα έπρεπε να μπορούμε να το προχωρήσουμε το θέμα, αλλά δεν θα δεσμευτούμε αν δεν μας δοθούν εγγυήσει ότι πράγματι υπάρχει βούληση συνεργασίας. Ξέρετε, θα μπορούσαμε να το είχαμε αποφύγει. Θα μπορούσαμε να είχαμε πει όχι, εξ αρχής αλλά ε, ξέρετε πολύ συχνά ότι η Ιρλανδία ε, φιλοδοξεί ε, έχει υπέρμετρες φιλοδοξίες και ενίοτε αυτό είναι πολύ καλό. Είμαστε υπέρμετρα φιλόδοξοι και παρά την κάμψη και την ύφεση στην Ευρώπη πιστεύουμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Εάν καταφέρουμε να συνεργαστούν όλοι θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο. Δεν σας υπόσχομαι τίποτα, δεν σας διαβεβαιώ ότι θα τα καταφέρουμε, ε, σας λέω μόνο ότι θα το προσπαθήσουμε. Από εκεί και πέρα, η απασχόληση δεν είναι ένα μόνο το ζήτημα της απασχόλησης. Η εντολή μου καλύπτει τέσσερις τομείς στην Ιρλανδία. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι πάρα πολλά, αλλά έτσι είναι η δουλειά μου έχω τις αναπηρίες, την ανισότητα, την τρίτη ηλικία και την ε, ψυχική υγεία. Και νομίζω ότι όλα αυτά ταιριάζουν αρκετά καλά μεταξύ τους. Αυτό πρέπει να το παραδεχθώ. Σε αυτούς τους τέσσερις τομείς, λοιπόν, το τελευταίο 1,5 χρόνο ε, προσπάθησα να καταλήξουμε σε μια συνολική κυβερνητική προσέγγιση για το πώς θα αντιμετωπίζουμε τα θέματα αυτά. Δηλαδή όταν ασχολούμαστε με την τρίτη ηλικία δεν μπορούμε να μιλούμε μόνο για την κοινωνική τους προστασία. Θα πρέπει να μιλήσουμε και για τη μεταφορά τους και για τη στέγασή τους και για την απασχόλησή τους ενδεχομένως. Όλα αυτά τα θέματα. Όταν μιλούμε λοιπόν για τις γυναίκες στην απασχόληση, δεν είναι μόνο το θέμα της απουσίας απασχόλησής τους. Υπάρχουν διάφορα άλλα ζητήματα με τις γυναίκες στην απασχόληση, άδεια μητρότητας, φροντίδα των παιδιών, ε, πρόσβαση στην εκπαίδευση. Όλα αυτά ε, συνδέονται μεταξύ τους. Μισθολογικές ανισότητες, το ίδιο ισχύει. Πρέπει να υιοθετήσουμε μια κοινή προσέγγιση πώς καταφέρνουν οι γυναίκες να εξοικονομήσουν χρόνο από την αγορά εργασίας για να είναι με τις οικογένειές τους και μετά να μπορούν να επανενταχθούν σε αυτή την αγορά εργασίας και πώς μπορούμε να, τα, να τις προστατεύσουμε σε αυτό. Η προσέγγιση μας οφείλει να είναι ρεαλιστική και συνεργατική. Να λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι... Ε, σε ορισμένες χώρες μέλη δεν έχει σημειωθεί τόση πρόοδος όσο σε άλλες χώρες μέλη αναφορικά με τα ζητήματα αυτά η βία κατά των γυναικών. Δεν έχω τόση ανοχή για το θέμα αυτό. Σε, σε άλλους τομείς ακολουθώ αυτή την προσέγγιση του λίγο-λίγο, βήμα-βήμα, σκαλί με σκαλή. Ε, στην βία κατά των γυναικών πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε μία άμεση λύση σαφέστατες δεσμεύσεις και δηλώσεις στα Ηνωμένα Έθνη, να δείξουμε τη σοβαρότητά μας. Εκεί δεν μπορούμε με το σταγονόμετρο. Πρέπει πράγματι εξ αρχής να ε, είμαστε παρόντες. Γιατί θεωρείτε, γιατί να θεωρείτε εντάξει, οκ, να είναι κανείς βίαιος εναντίον των γυναικών. Δεν μπορεί να θεωρείται κάτι τέτοιο. Αυτό πρέπει να το ε, πούμε ξεκάθαρα, να το δηλώσουμε απερίφραστα. Και το EPO, η Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας δηλαδή, ε, είναι μια εγγύηση. Δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά είναι ένα πρακτικό βήμα που θα βοηθήσει κατά πολύ ε, την προστασία των γυναικών. Δεν θα χρειαστεί δηλαδή ε, μία γυναίκα συνεχώς να φοβάται, ε, μία γυναίκα συνεχώς να νιώθει ανησυχία όταν μετακινείται είτε για να πάει στο χώρο εργασίας της, είτε για να είναι με τα παιδιά της. Δεν θα πρέπει να ξεκινά τη διαδικασία ξανά και ξανά. Είναι ένα από τα πρακτικά βήματα η Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το κάνει αυτό πάρα πολύ καλά. Αναγνωρίζουμε όλοι ότι πρέπει να συνεργαστούμε για τα ζητήματα αυτά, γιατί τελικά ο κόσμος μας είναι πολύ μικρός πλέον. Άρα χρειάζεται συνεργασία όλων μας. Νομίζω ότι όλοι έχουμε ακριβώς την ίδια άποψη για το θέμα της βίας εναντίον των γυναικών. Είμαστε πολύ σοβαροί στις προσεγγίσεις μας ακροτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων. Έχουμε πανίσχυρη νομοθεσία στην Ιρλανδία για το θέμα αυτό. Δεν είμαι καθόλου βεβαία ότι η Προεδρία, ο Πρόεδρος ε, της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνει αυτά που του ζητάτε. Ωστόσο, σας διαβεβαιώ ότι με απόλυτη σοβαρότητα αντιμετωπίζουμε τα θέματα ε, που έχουν να κάνουν με τη βία εναντίον των γυναικών, η οποία είναι μία από τις πιο ιδεχθείς μορφές βίας. Και θα πρέπει το θέμα αυτό να είναι πάντοτε στο προσκήνιο, να δηλώνεται απερίφραστα πόσο απαράδεκτη είναι αυτή η μορφή ιδεχθούς βίας. Και νομίζω ότι το Συμβούλιο αυτό το έχει διακηρύξει απερίφραστα. Ως προς τις συντάξεις, είναι ένα ζήτημα για όλη την Ευρώπη. Μας αφορά όλους. Πρέπει να το εξετάζουμε προσεκτικά. Οφείλουμε να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες καθώς γερνούν, να παραμείνουν στο χώρο εργασίας, να παραμείνουν ενεργά μέρη της οικονομίας. Είναι αναπόσπαστο μέρος αυτό ε, του, της λύσης του προβλήματος του συνταξιοδοτικού. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο το πρόγραμμα για την ε, ηθαγένεια, για τους πολίτες, για τα δικαιώματα, κατά πόσο θα προχωρήσουμε εκεί. γίνεται κεντρική διαπραγμάτευση για τα του προϋπολογισμού. Εμείς θα το στηρίξουμε πολύ αυτό το πρόγραμμα και θα υπάρξει πρόοδος γιατί πρέπει να υπάρξει τελικά. Τα ζητήματα που συζητούμε σήμερα είναι ζητήματα που μας αφορούν όλους. Δεν αφορούν μόνο την δική σας επιτροπή, αλλά θα έπρεπε να αφορούν και αφορούν όλες τις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. στηρίζουμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όποτε αυτές ε, προκύπτουν πριν από τις δικές μας και πάντοτε θα ε, παρουσιάζουμε την άποψή μας για το θέμα αυτό. Σας μίλησα ήδη για το CSW, για το καθεστώς των γυναικών, την ε, Σχετική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών. Θα έχουμε πολύ σύντομα μια ισχυρή ευρωπαϊκή θέση για τα θέματα αυτά πρέπει τα Ηνωμένα Έθνη να είναι όσο το δυνατόν πιο ισχυρά ώστε να ε, επιτύχουν τους στόχους τους και εμείς πρέπει να τους βοηθήσουμε σε αυτό. Για τη βία εναντίον των γυναικών μίλησα, για την οδηγία κατά των διακρίσεων δεν μπορώ να σας, υποσχεθώ ότι θα ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες κατά τη διάρκεια της ε, ε, Προεδρίας μας. Θα δώσουμε προτεραιότητα στον φάκελο αυτό και ειδικότερα ως προς τις αναπηρίες, ε, τα άτομα με αναπηρίες ε, ε, για τα οποία έχω αρμοδιότητα επίσης, ούτως ώστε να προστατευτούν οι άνθρωποι αυτοί από τις διακρίσεις που όλοι γνωρίζουμε ότι υφίστανται. Τώρα, ο αντίκτυπος της κρίσης στις γυναίκες της Ιρλανδίας. Με ρωτήσατε γι' αυτό. Να σας πω ότι και εδώ πιστεύω ότι το σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι προστατεύουμε το πληθυσμό στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Προστατεύουμε το λαό στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στο βαθμό του δυνατού. Χωρίς να εμπλεκόμαστε τόσο πολύ στην κρίση ώστε να ξεχνούμε τις απαραίτητες δομές που θα βοηθήσουν τις χώρες να βγουν από την κρίση. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια της κρίσης πρέπει να έχουμε τις κλασικές δομές που στηρίζουν μια κοινωνία, ώστε όταν μια κοινωνία βγει από την κρίση να μπορεί να στηριχθεί πάλι σε αυτές τις δομές και υποδομές τελικά. Δουλειά μας είναι να αξιολογούμε, να διασφαλίζουμε τελικά ε, ότι όταν η, η χώρα βγει από την κρίση θα μπορεί να σταθεί πάνω σε γερά θεμέλια. Ε, δεν σημαίνει ότι ε, όλα πρέπει να γίνουν τώρα. Ορισμένα πράγματα μπορεί να μην μπορούν να γίνουν λόγω της οικονομικής ύφεση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνουν στο μέλλον. Βεβαίως και θα μπορούν να γίνουν στο μέλλον. Ε, αυτά προς το παρόν σας ευχαριστώ πολύ. Θα ολοκληρώσω στα σουηδικά. Θα συνοψίσω στα Σουηδικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολλές οι ερωτήσεις, πολλές οι παρατηρήσεις. Ε, όπως βλέπετε όμως ενδιαφέρεται πάρα πολύ η ε, Επιτροπή μας για τα θέματα αυτά. Προσβλέπουμε λοιπόν στην Προεδρία σας ε, και όσον αφορά την επίσκεψη ε, στη Νέα Υόρκη, στο CSW θα είμαστε παρόντες. Εγώ και τέσσερα άλλα μέλη της Επιτροπής μας θα είμαστε παρόντες. Υπάρχει λοιπόν ε, πολύ καλή δυνατότητα συνεργασίας εκεί. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μπόρεσες να έρθεις εδώ σήμερα. Ευχαριστώ και πάλι και καλή επιτυχία.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 to vote. So please take your seat. Να ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες, παρακαλώ καθίστε. You want to speak, you are extremely free to do. Αν θέλετε να πάρετε, αν θέλετε να μιλήσετε, πολύ ευχαρίστως να συνεχίσετε, αλλά έξω από την αίθουσα. Ωραία. Θα μιλήσω σου ειδικά. Περνάμε στις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Έχουμε την απαλλαγή του 2011 Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων. Να ρωτήσω αν η συγγήτρια η κυρία Κλειβέτη θέλει να πάρει το λόγο. Thank you very much, uh, President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω είναι σημαντική έκθεση αυτή. Με ακούτε? Τι θέλετε να μιλήσω ρουμανικά? Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι η έκθεση να ψηφιστεί όπως την πρότεινα. Διότι θα είναι ένα σημαντικό μήνυμα από την Επιτροπή μας να ενθαρρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει μέρημνα για την χρηματοδότηση της, του θέματος της ισότητα των φίλων. Θα είναι ένα σημαντικό μήνυμα. Ωραία, περνάμε στην ε, ψηφοφορία. Τροπολογία 5 υπέρ, κατά, αποχές. Απορρίπτεται από ό,τι βλέπω. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η εννέα έχει αποσυρθεί. Έχουμε την τελική ψηφοφορία, η ηλεκτρονική, ε, αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Σημείο 13. Απαλλαγή 2011. Γενικό Προπολογισμό Ευρωπαϊκή Ένωση. Τμήμα 3. Επιτροπή. Μία τροπολογία έχουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Έχουμε την τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχή τη ψηφοφορία. Λήξη τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Προχωράμε στο 14. Εξάλληψη και πρόληψη όλων των μορφών βία κατά των γυναικών και των κορισιών εν ώψη της 57ης Επιτροπής του ΟΗΕ για το καθεστώ των γυναικών, CSW. Ε, ξεκινάμε πρώτα με μια προφορική ερώτηση. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω πρέπει να την ελέγξουμε. Τροπολογία 1, ελέγχουμε υπέρ. Ε, μάλλον, ε, συγγνώμη, ψηφίζουμε. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4, υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 6 έχει αποσυρθεί. Η τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 έχει αποσυρθεί. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έχουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία, αρχή της ψηφοφορίας για το ψήφισμα, λήξη της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Έχουμε πρόταση ψηφίσματος, τροπολογία 9, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 10, υπέρ, κατά,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 Αρχή της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Χωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Πολύ δύσκολο να διακρίνω. Να το ελέγξουμε. Το δεύτερο μέρος χωριστή, της χωριστής ψηφοφορίας, αρχή της ψηφοφορίας. The vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία. Υπάρχει αντίρρηση στην υποβολή της προφορικής τροπολογίας. Όχι, ωραία, ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Έχουμε και άλλη προφορική τροπολογία. Έχει κανείς αντίρρηση στην υποβολή αυτής της προφορικής τροπολογίας. Ωραία, ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε πάνω στο σύνολο του ψηφίσματος αρχή τη ψηφοφορία. Λήξη τη. ψηφοφορία. Όχι, οι σοσιαλδημοκράτες δεν ψήφισαν. Ε, συγγνώμη, μάλλον οι σοσιαλδημοκράτε έχουν μία ψήφο παραπάνω, αλλά ούτω ή άλλω βλέπω ότι δεν παίζει ρόλο. Να ξαναψηφίσουμε. Οι σοσιαλιστέ και οι δημοκράτε έχουν μία ψήφο παραπάνω. Ε, επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία αρχή τη ψηφοφορία. Ελάτε, λήξη τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Και τέλος, σημείο 15, εκπόνηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου όσον αφορά τη χρηματοδότηση της συνεργασία Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού κλπ. Να ρωτήσω μήπως ε, η εισηγήτρια θέλει να πάρει το λόγο, όχι. Ωραία, αρχίζουμε με την τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ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 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται. Να ελέγξουμε την 27. Αρχή της ψηφοφορίας. The vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. 27 απορρίπτεται. Φορά τα γυαλιά μου. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31. Χωριστή ψηφοφορία σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές. Πολύ δύσκολο να διακρίνουμε. Ελέγχουμε λοιπόν το πρώτο μέρος, αρχή τη ψηφοφορίας. And the vote is closed. Λήξη της ψηφοφορίας. Εκρίνεται. Το δεύτερο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το τρίτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να ελέγξουμε τι δύο πρώτε μετά θα ρωτήσω πώ μπορούμε να τι πάρουμε όλε μαζί. Τροπολογία 32, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 33, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και κατόπιν ρωτώ, μπορούμε να ψηφίσουμε όλες τις υπόλοιπες μαζί. Δεν έχει κανείς αντίρρηση, ωραία. Α, υπάρχει αντίρρηση.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 Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται σαφώς. Σας ευχαριστώ πολύ. <laughs> Θα ξεκινήσουμε πολύ σύντομα τη συνεδρίαση, αλλά πρέπει να περιμένουμε δύο-τρία λεπτά. Και θα συνεχίσουμε.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

Eh, Μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Και περνάμε στο σημείο 16. Εκπαιδευτική και επαγγελματική κινητικότητα των γυναικών στην Ευρώπη. Έχουμε το πολύ μισή ώρα στη διάθεσή μας. Θα ήθελα λοιπόν πρώτα να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια την κυρία Ρονζούλη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια σύντομη εισαγωγή και μετά θα περάσω στις λεπτομέρειες του περιεχομένου η Ευρώπη τα ερχόμενα χρόνια καλείται να αντιμετωπίσει σημαντικέ προκλήσει επειδή η αγορά εργασία ανοίγει όλο ένα και περισσότερο και υπάρχει μεγαλύτερη πρόσβαση. Βεβαίω παραμένουν φραγμοί για την κινητικότητα των εργαζομένων σήμερα μεταξύ των κρατών μελών. Υπάρχουν ανισότητε, επίση ελλείψει στι γλωσσικέ γνώσει. οι ευνοϊκέ συνθήκε για τη συμφιλίωση επαγγελματικού και οικογενειακού βίου ακόμη δεν είναι πρόσφορε και χρειάζεται ενημέρωση των εθνικών νομοθεσιών για ζητήματα πρόνοιας. Η πρόσβαση στις πληροφορίες για την διασυνοριακή κινητικότητα επίσης είναι ελλειπής και χαμηλής ποιότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα ερχόμενα χρόνια πρέπει να αναλάβει τη δέσμευση, να ευνοήσει και να προωθήσει την επαγγελματική κινητικότητα. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα το πετύχουμε μόνο με την ενημέρωση των σημερινών, των ισχυόντων συστημάτων κατάρτιση και εκπαίδευση, δίνοντα μεγαλύτερη σημασία στι ε, μεγαλύτερε απαιτήσει τη αγορά εργασία και δίνοντα τη δυνατότητα τη διαρκού μάθηση, καθώ και με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Θυμίζουμε ότι πρώτος στόχος της στρατηγικής της Ευρώπης το 2020 είναι να φτάσει στο 75% το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών και των ανδρών στην ηλικία 20 έως 64 έτη είναι σημαντικό ένα ένα μεγαλύτερο ποσοστό ε, προσώπων να μπορούν να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας όπως για τις γυναίκες που προσωρινά μπορεί να βγουν από τον επαγγελματικό βίο λόγω της μητρότητας. Η απασχόληση θα πρέπει να έχει ευνοϊκότερες συνθήκες για, τους, για τις γυναίκες. Επίσης, την ανάπτυξη θα την προωθήσουμε μόνον εφόσον δώσουμε κίνητρα για επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο και την παραγωγικότητα των γυναικών. Βεβαίως, εδώ υπάρχει θέμα με τους ανθρώπινους πόρους. Το περιεχόμενο της έκθεσης έχει χωριστεί σε αιτιολογικές σκέψεις και άρθρα. Προφανώς, στις αιτιολογικές σκέψεις υπογραμμίζεται το δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών να παραμένουν και να εργάζονται σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέραν της δικής τους, η συμβολή της επαγγελματικής κινητικότητας στην ε, τόνωση του συναισθήματος ε, του ανήκειν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, σημαντική. Από την άλλη, η οικονομική κρίση έχει πλήξει πολλές επαγγελματικές κατηγορίες στην αγορά εργασίας, ιδίως τι γυναίκες. Βεβαίω υπάρχει ακόμη απόκληση μεταξύ των δύο στην αγορά ε, εργασίας, οπότε εδώ πρέπει να δοθεί έμφαση στη διαρκή μάθηση και τη συμφιλίωση του επαγγελματικού με τον οικογενειακό βίο, καθώς και την καλύτερη πρόσβαση των γυναικών στην αγορά εργασίας. Στα άρθρα δίνεται έμφαση στην προώθηση της ισότητας των φύλων, στις ίσες ευκαιρίες, στην καταπολέμηση κάθε μορφής εκμετάλλευσης ε, στην αγορά εργασίας, στην προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών ε, ως προς την κινητικότητα την επαγγελματική μέσω των εθνικών νομοθεσιών ενώ επιπλέον υπογραμμίζεται ότι συχνά οι γυναίκες μετακινούνται στο εξωτερικό για να αναλάβουν επαγγελματικά καθήκοντα που έχουν να κάνουν με φροντίδα ηλικιωμένων ή παιδιών. Αυτές προσλαμβάνονται χωρίς κανένα συμβόλαιο σύμβαση ή ακόμα χειρότερα δουλεύουν λαθρέα, παράνομα, χωρίς καμία ε, προστασία ή εγγύηση στις γυναίκες πολλές φορές προσφέρονται θέσεις εργασίας χαμηλού επίπεδου, όχι μόνο από την πλευρά των αρμοδιοτήτων που καλούνται να ασκήσουν, αλλά και από πλευρά κύρους ή αμοιβής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη καλούνται να παρακολουθήσουν την παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών στην αγορά εργασία. Προφανώ πρέπει να παρακολουθούν τι καταστάσει που μπορεί να δημιουργούνται και πρέπει να ενισχυθεί η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της διακριτικής μεταχείρισης, είτε είναι έμεση είτε άμεση, κατά των αλλοδαπών εργαζομένων. Επίσης θα πρέπει να δημιουργηθούν εθνικά σημεία επαφής για τις ανεξάρτητες εργαζόμενες ώστε να υπάρχει ανταλλαγή στοιχείων, ένα είδος πλατφόρμας. Επίσης διαφάνεια για να αντιμετωπιστούν οι μισθολογικές ανισότητες βάσει των φύλου και έκκληση προς τα κράτη-μέλη να προβλέψουν διαρθρώσεις και υπηρεσίες για τα παιδιά στην περίπτωση που ένας εργαζόμενος αναγκαστεί να μεταναστεύσει μαζί με την οικογένειά του. Θα πρέπει να εξαλειφθούν οι φραγμοί κατά της επαγγελματικής κινητικότητας μέσω της προσφοράς κατάλληλων υπηρεσιών όπως γλωσσικά μαθήματα. Ένας φραγμός που απαντάται συχνά. Δεν είναι όμως και το δυσκολότερο να ξεπεραστεί ως εμπόδιο. Επίσης θα πρέπει να προωθηθεί η διαρκής μάθηση και η επαγγελματική κινητικότητα, να υποστηριχθεί το πρόγραμμα Εράσμους και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να παράσχουν πρόσθετη βοήθεια στις άγαμες μητέρες ή να αυξήσουν το επίπεδο των ε, γυναικών που μετακινούνται στο εξωτερικό με διαβίου μάθησης προγράμματα. Να θυμίσω εδώ ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι στις 29 Ιανουαρίου στις 12 το μεσημέρι. Οι τροπολογίες θα συζητηθούν 18-19 Φεβρουαρίου λίγο πολύ τι τροπολογίε θα τι συζητήσουμε στι 20 Μαρτίου. Την ψηφοφορία στην Επιτροπή Γυναικών, αν δεν αλλάξει το χρονοδιάγραμμα, θα την έχουμε 22-23 ε, Απριλίου και θα περάσει στην Ολομέλεια του Στρασβούργου τον Μάιο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω πρώτο λόγο στην κυρία Νιβεντάλοβα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά. Λίγα πράγματα μπορώ να προσθέσω. Δώσατε έμφαση στα εμπόδια που θα πρέπει να καταρριφθούν. Και καλός. Πολύ καλός. Πολλά είναι τα εμπόδια στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας και πολλά είναι τα εμπόδια μετά, κατά τη διάρκεια της εργασίας δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην ε, υψηλότερη εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών. Είναι κάτι που πρέπει να υποστηρίξουμε. Το τονίζεται αυτό. Τονίζεται και την ανάγκη στήριξης των γυναικών κατά τη διάρκεια της άδεια μητρότητας. Μου αρέσει πολύ το άρθρο 9 όπου λέτε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να στηρίζουν τους άντρες ή τις γυναίκες που είναι μαζί με τον ή την σύντροφό τους και τα παιδιά τους. Θα πρέπει να προσφέρονται υπηρεσίες φύλαξης και φροντίδας των παιδιών σε πολύ μικρή βρεφιακή νηπιακή ηλικία. Μου αρέσει το άρθρο 10 που αναφέρεται τα μαθήματα γλώσσας για τη συζύγους ή τους συζύγους που πηγαίνουν με τον σύντροφό τους όταν αυτός ή αυτή βρίσκει μια θέση, μια θέση απασχόλησης στο εξωτερικό, ώστε να ενταχθούν καλύτερα στην κοινωνία, στον τόπο υποδοχής, στο νέο του σπιτικό. Μου αρέσουν αυτές οι διατυπώσεις, θα τις στηρίξω. Θα πρέπει επίσης να υποστηρίξουμε τις νέες τάσεις στην κινητικότητα. Να αναφέρουμε το γεγονός ότι όλο και περισσότερες γυναίκες πηγαίνουν στο εξωτερικό για να δουλέψουν οι ίδιες. Δεν ακολουθούν τους συζύγους τους. Νέες γυναίκες, αλλά και μεγαλύτερης ηλικία γυναίκες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης πηγαίνουν στο εξωτερικό για να εργαστούν και θα πρέπει να τις υποστηρίξουμε. Να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να έχουν πρόσβαση στα συστήματα υγείας. Οι γυναίκες που πηγαίνουν στο εξωτερικό για να εργαστούν προσφέροντας φροντίδα είτε σε παιδιά είτε σε ηλικιωμένους μεταξύ άλλων. Όλα αυτά θα πρέπει να αναφερθούν, θα πρέπει να τα υπογραμμίσουμε και να τα διεκδικήσουμε. Αναφερθήκατε και σε κάτι το εξαιρετικά σημαντικό, την εκπαιδευτική κινητικότητα. Δεν θέλω να περιοριστώ στο πρόγραμμα Εράσμος που αναφέρεται σε μία από τις παραγράφους. Έχουμε και το Κομένιος, έχουμε και το Κρούμβιχ. Δεν μιλούμε μόνο για την κινητικότητα των φοιτητών του Πανεπιστημίου, μιλούμε και για την κινητικότητα των καθηγητών. Χρειάζονται οι καθηγητές τέτοιου είδους εμπειρίες. Ίσως πρέπει να αναφέρετε πολλά προγράμματα, να μην περιοριστείτε μόνο στο Εράσμος. Και μια και μιλούμε για αυτό το θέμα, καλό θα ήταν να αναφερθεί και ένα καινούριο πρόγραμμα, το οποίο τελικά θα περιλάβει όλα αυτά. Ο τίτλος εργασίας για την Ευρώπη. Να μιλήσουμε δηλαδή για αυτό το πρόγραμμα κινητικότητας για την επόμενη περίοδο. να ενημερώσουμε την έκθεση αυτή με τα καινούργια δεδομένα. Και κάτι που αναφέραμε και χθες, το 60% των πτυχιούχων πανεπιστημίου είναι γυναίκες. Και πρέπει να υπερασπιστούμε το δικαίωμα όλων στην πρόσβαση ε, στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Αυτό ναι και καλώς το αναφέρεται. Θα πρέπει όμως να μεριμνήσουμε ότι τελικά οι πτυχιούχοι μπορούν να βρουν δουλειά, μπορούν να βρουν μια θέση στη ζωή και στην κοινωνία και μετά το πανεπιστήμιο. Καλό θα ήταν ενδεχομένως να αναφέρουμε το γεγονός ότι θέλουμε να στηρίξουμε τις νέες πτυχιούχους, γυναίκες πτυχιούχους, άλλωστε το 60% των πτυχιούχων είναι γυναίκες όπως σας είπα, το 40% εξ αυτών βρίσκουν θέση απασχόλησης και θα πρέπει να το αναφέρουμε στην έκθεση. Και κάτι που είπα και χθες. Όταν μιλούμε για την άδεια μητρότητας, ενδεχομένως θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για το μοίρασμα των δουλειών, job sharing. Ε, ίσως τελικά παρανοήθηκα χθες, δεν έγινε αντιληπτή. Ε, έχουμε μερική απασχόληση και θα μπορούσαν οι γυναίκες που είναι σε άδεια μητρότητα να την κάνουν μισή-μισή με κάποια γυναίκα τρίτη ηλικία που ενδεχομένω έχει πάρει σύνταξη. Και αυτό να είναι ένα εργαλείο που να μπορούν να αξιοποιούν και οι άνδρες. Να δούμε πώς θα το διατυπώσουμε, αλλά να υπάρχουν τέτοιου είδους εργαλεία ευελιξίας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας και συγχαρητήρια για τη δουλειά σας. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ η κυρία Μπλίκοβιτσια. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Καταρχήν, ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, κυρία Ρονζούλη για την εξαιρετική της έκθεση. Συμφωνώ ότι ε, γίνονται διακρίσεις λόγω φύλου στην επαγγελματική ζωή που έχουν σημαντικές επιπτώσεις για τις γυναίκες όσον αφορά τη σταδιοδρομία τους, την αμοιβή τους, και την ικανοποίηση ε, από τη δουλειά τους. Ε, θα ήθελα να κάνω κάποιε παρατηρήσει για την έκθεση αυτή. Πέρα από την εκπαίδευση ε, και ένταξη και απασχόληση των γυναικών, στην έκθεση αυτή θα πρέπει να μιλάμε και για την υγεία, την φτώχεια, την ψαλίδα στι αμοιβέ και τον ρόλο τους στην λήψη αποφάσεων. προτείνω όσον αφορά τα θέματα αυτά να αναφερθούμε σε διάφορε ηλικιακέ ομάδε γυναικών, διότι κάθε ηλικιακή ομάδα έχει τα ιδιαίτερα προβλήματά τη. Ε, δεύτερον, θα πρέπει να παίξουμε περισσότερο θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη προσοχή στην ένταξη των γυναικών ε, στην ε, αγορά εργασία. Ε, να είναι δυνατόν για τι γυναίκε να αλλάξουν τι δεξιότητέ του, να αναπτύξουν δεξιότητε, να βρουν δουλειέ υψηλή ποιότητα σύμφωνα με τι δεξιότητές τους και σήμερα οι γυναίκες έχουν όλο και καλύτερη εκπαίδευση, κάτι που ε, αυξάνει το ποσοστό απασχόλησης τους, ε, αλλά η δυσκολία συνδυασμού οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής αποτελεί τον βασικό ρόλο που ε, οι περισσότερες γυναίκες έχουν δουλειές χαμηλής βαθμίδας. είμαι σκιώδης συγητή στην Επιτροπή Απασχόλησης ε, και νομίζω ότι αν συνεργαστούμε θα μπορέσουμε να προωθήσουμε τις ε, ε, ευκαιρίες των γυναικών στην εκπαίδευση και την επαγγελματική ζωή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ρωτήσω αν κάποιος από την Επιτροπή θα θέλει να πάρει το λόγο. Όχι. Ωραία. Α, παρακαλώ. να ζητήσω συγγνώμη γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπόρεσε να στείλει πρόσωπο. <laughs> δεν υπάρχει πρόβλημα. Ε, I to... Να δώσω το λόγο πάλι στην κυρία Ρουτσούλη, παρακαλώ. Εάν θέλετε να κάνετε κάποιες τελικές παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Όχι, απλώς να ευχαριστήσω τις συναδέλφους Για, τα για τις μισθολογικές διαφορές νομίζω αναλύεται αρκετά στην έκθεση. Απλώς να ευχαριστήσω και τη συνάδελφο της οποίας δεν μπορώ να καταφέρω να προφέρω το όνομα σωστά. Μπλινκεβι Κούτε. Όντως έχει να κάνει και με την ηλικία αυτό. Κάθε ηλικιακή ομάδα δεν έχει απλώς διαφορετικές ε, ε, διαφορετικά χαρακτηριστικά αλλά και ανάγκες. Την ευχαριστώ λοιπόν και περιμένω τις τροπολογίες των συναδέλφων. Ελπίζω ότι θα συνεργαστούμε αρμονικά. Σας ευχαριστούμε. Και τώρα να σας δώσω απλώς το χρονοδιάγραμμα. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 28 Ιανουαρίου στις 5 το απόγευμα. Το θέμα θα συζητηθεί 19, 18 ή 19 Φεβρουαρίου και θα ψηφίσουμε 22-23 Απριλίου. Στην Ολομέλεια μάλλον θα περάσει το θέμα το Μάιο. Ολοκληρώνουμε και με το θέμα αυτό και περνάμε στο επόμενο σημείο που θα είναι το 17. Σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και δικαιώματα. Ακριβώς το απόγευμα για το θέμα αυτό θα έχουμε ακρόαση. Ακρόαση 3 έως 6.30 σήμερα. Ελπίζω να είναι ενδιαφέροντα τα αποτελέσματα. Μια έκθεση που θα δούμε αργότερα μέσα στη χρονιά. Και βεβαίως η ακρόαση έχει να κάνει με το θέμα αυτό. Να πω ότι οι προσεχείς μας συνεδριάσεις, υπό το σημείο 18, προβλέπονται 18 Φεβρουαρίου 3 με 6.30 και 19 Φεβρουαρίου 9 με 12.30. Έχουμε ολοκληρώσει με την ε, συνεδρίασή μας. Ευχαριστώ.